started. Συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε αυτή τη σημαντική ακρόαση. Είμαι ευτυχής που οι δυο μας επιτροπές, ε, η, αρμόδια για τις υποθέσεις των γυναικών και η ΛΥΜΠΕ, ε, ναι, μη στεναχωριέστε, θα έρθουν κι άλλοι. Σίγουρα βλέπουν και διάφοροι από το διαδίκτυο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η ακρόαση και δείχνει πως οι δυο μας επιτροπές συνεργάζονται στενά. Και... Είμαι ευτυχής που αυτή η αγαστή συνεργασία συνεχίζεται. Και έχουμε εδώ τον συμπρόεδρο Πιμέντα Λόπες, που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Γυναικών. Σε ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Συνάδελφοι, θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια εισήγηση για τη σημερινή ακρόαση. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Να ακούσουμε πρώτα τους ε, προσκεκλημένους μας. Ε, να δούμε λοιπόν τι συζητάμε σήμερα. Έχουμε να μιλήσουμε για το πολύ σημαντικό θέμα του εμπορίου παιδιών και γυναικών στο πλαίσιο της μετανάστευσης που φαίνεται να είναι ένα ζήτημα που όλοι γνωρίζουμε, όλοι μας έχουμε άποψη γιατί πρόκειται για την δουλεία των καιρών μας αλλά σήμερα θέλουμε να μπούμε πιο εις βάθος και να δώσουμε απαντήσεις νομοθετικού τύπου ώστε να αναπτύξουμε πιο στοχοθετημένη απάντηση. Βεβαίω ε, έχουμε συζητήσει την ε, εμπορία ανθρώπων ε, επανελειμμένα και στις δύο Ε, σήμερα θα μιλήσουμε για την οπτική γωνία της εμπορίας μέσα στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Οι διακινητές, οι λαθρέμποροι εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ε, ε, κατάσταση και εφόσον δεν υπάρχουν νόμοι μεσοδοί για να φτάσουν οι μετανάστες από τρίτες χώρες ε, εκμεταλλεύονται. Δεν υπάρχουν νόμοι μεσοδοί αυτή τη στιγμή. Και αν υπάρχουν, είναι περισσότερο αφορούν εθνικές περιπτώσεις και όχι ευρωπαϊκές. Έχουμε αυτό το πρόβλημα, είναι όλοι στα όρια της νομιμότητας αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να μεταναστεύσουν και καταλήγουν σε καταστάσεις όπου η ακεραιότητά τους και η ελευθερία τους κινδυνεύουν. Έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές επικίνδυνες καταστάσεις και Έχουμε τον δρόμο του Αγκαντές προς τη Λιβύη και προσπαθούμε να απαντήσουμε από τις πιο επικίνδυνες καταστάσεις. Εγώ πρόσφατα επισκέφθηκα τη Λιβύη και είδα τους καταβλισμούς προσφύγων, είδα ε, επίσης τις εγκαταστάσεις του IOM στο Αγκαντέζ και ε, τακτικά ε, γίνονται καταχρήσεις και βιασμοί σε αυτούς τους, τους δρόμους της μετανάστευσης. Και στην Επιτροπή μας ε, λοιπόν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να ε, απαντήσουμε σε αυτό το ανθρωπιστικό βήμα και με στρατηγικό τρόπο, σε αυτό το πρόβλημα μάλλον με στρατηγικό τρόπο. Έχουμε λοιπόν ε, να δούμε την κατάσταση των γυναικών και των παιδιών και φυσικά αυτό εξηγεί και την συσχέτιση των δυο μας επιτροπών. Να δώσω σύντομα το λόγο και στον Συμπροεδρό, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Γυναικών, τον κύριο Ζωάου Πιμέντα Λόπες, που θα κάνει μια σύντομη εισήγηση και θα παρουσιάσει τους ομιλητές. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ που που υπάρχει αυτή η συνεργασία ανάμεσα στις δύο επιτροπές όπως είπατε. Πράγματι είχα την ευκαιρία για να προετοιμάσω δύο λόγια εισαγωγικά για αυτήν εδώ την ακρόαση και μπόρεσα να δω κάποιες από τις συμβολές που έχει κάνει η Επιτροπή των Γυναικών στο ιδιαίτερο πλαίσιο της μετανάστευσης και στο συγκεκριμένο πλαίσιο που σήμερα θα συζητήσουμε της εμπορίας ανθρώπων ανθρώπων, ιδιαίτερα παιδιών και γυναικών. Ήταν εύκολο να δούμε την άμεση συμβολή της Επιτροπής Γυναικών. Ε, έχει ενημερώσει για τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν τα παιδιά και οι γυναίκες, το θέμα των αναγκών της, ε, των γυναικών, τα θύματα οι ιδιαιτερότητες των ανήπανδρων μητερών, των ε, πολύ νέων μητερών, τα προβλήματα των θυμάτων σωματικής ή ψυχολογικής βίας, τα θέματα των υποδομών ε, και της έλλειψης ε, υποδομών οι οποίες να είναι προσαρμοσμένες στην κουλτούρα, ε, την νοοτροπία των θυμάτων. Αλλά βέβαια οριζόντια σε όλα τα κείμενα που έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε μιλήσει και για το θέμα του φύλου και αναπόφευκτα όλα αυτά ε, διαποτίζονται από την ε, μεταναστευτική μας πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν υπάρχουν εγγύησεις και δεν, ε, ο τρόπος με τον οποίο ασκείται αυτή η πολιτική δεν δίνει λύσεις. Έχουμε διάφορα ψηφίσματα στο Κοινοβούλιο που αφορούν ακριβώς την ανάγκη ε, νόμιμων και ασφαλών οδών ώστε να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε και να καταπολεμήσουμε το εμπόριο ανθρώπων. Και αυτό συνδέεται και με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το θέμα του εμπορίου ανθρώπων και η Ε, ο εντοπισμός των ιδιαίτερη της ιδιαίτερης κατάστασης των κοριτσιών, των ανήπανδρων μητέρων και των γυναικών ε, ευρύτερα στο πλαίσιο της μετανάστευσης δίνει, έχει μάλλον ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γι' αυτό και το τονίζουμε ε, στο πλαίσιο του εμπορίου ανθρώπων. Αυτό το εμπόριο θέλει να τροφοδοτήσει νέες μορφές ε, σκλαβιάς και εκμετάλλευσης στο 21ο αιώνα σε τομείς όπως η γεωργία ή οι, οι, ε, οικοδομές. Η εμπορία όμως γυναικών είναι, έχει ακόμα πιο βίο χαρακτήρα γιατί πρόκειται για τροφοδότηση νοσηρών, νοσηρού εμπορίου εμπορίου όπως αυτό της ε, ε, εκπόρνευσης γυναικών. Υπάρχει δηλαδή και κοινωνικό ζήτημα εδώ ε, και γι' αυτό και θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στη σημερινή συζήτηση να δούμε, να ακούσουμε μάλλον πώς οι ομιλητές που θα παρέμβουν στις δύο συνεδρίες θα μιλήσουν για το θέμα του εμπορίου γυναικών και παιδιών τόσο σε σχέση με τις άμεσες απαντήσεις που είναι δυνατόν να δώσουν για την ε, εμπορία αλλά και θίγοντας αυτά τα θέματα που φαίνεται να να είναι παράπλευρα, ωστόσο είναι άμεσα συνδεδεμένα, αλληλένδετα με την εμπορία παιδιών και γυναικών, αλλά και με την μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης, αλλά και τις πολιτικές της Ένωσης και των κρατών μελών στην καταπολέμηση της ε, ε γυναικών και παιδιών και ε, ιδιαίτερης εκμετάλλευσης ε, της σεξουαλικής, της έκδοσης παιδιών και γυναικών. ο κύριος Μωράης. Μπορείτε να παρουσιάσετε τώρα τους ομιλητές που θα μας παρουσιάσουν τις ομιλίες τους. Να αναφέρω μόνο ότι θα πρέπει να αποχωρήσω στις 11 για ε, μια συνεδρίαση προανελημένη υποχρέωση δεν θέλω, δεν θέλω να το κλάβετε ως έλλειψη σεβασμού ή ενδιαφέροντος να ευχαριστήσω και τις δύο γραμματείες που συνδιοργάνωσαν ε, την σημερινή ακρόαση για το ότι προσκαλέσατε τόσο εξαιρετικούς ομιλητές. Θέλω επίσης να αναφέρω ότι αν και δεν βλέπετε πολλούς βουλευτές παρόντες, πολλοί κόσμος παρακολουθεί στο διαδίκτυο όπου αναμεταδίδεται ζωντανά η συνεδρίαση. Κάποιοι από τους συναδέλφους έχουν δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για αυτά τα θέματα Απλά ήθελα αυτό να το πω πριν να αποχωρήσω. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα τώρα. Λοιπόν, θα σταματήσω να μιλάω εγώ. Ε, και ε, μπορείτε να παρουσιάσετε τους ομιλητές. Μάλιστα. Θα, δώσουμε, θα ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη συνεδρία πρόληψη και προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Θα ακούσουμε πρώτα τις διάφορες προοπτικές και τις διάφορες απόψεις. Πρώτη παρέμβαση είναι η θεσμική προσέγγιση του IOM από πλευράς του κυρίου Ευγένιο Αμπρόζη που θα μας παρουσιάσει μια μελέτη που εκπώνησε η UNICEF. Μετά έχουμε μια πιο ακαδημαϊκή προοπτική μέσα από την οπτική, την ανθρωπολογική, που δεν, ε, ε, ε, δεν αναλύεται πάντοτε από τον κύριο Μιχάλκο και τέλος θα πάρει το λόγο η κυρία Κατίζ για να μας δώσει την εικόνα επιτόπου ε, λάβετε υπόψη ότι εργάζεται με μια μη κυβερνητική οργάνωση που στηρίζει τις ε, νιγηριανές γυναίκες θύματα της ε, εμπορίας ανθρώπων. Ο κάθε ομιλητής έχει 8 λεπτά, πρώτος ο κύριος Αμπρόζη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να απευθύνω το λόγο εδώ στην Επιτροπή ε, σε αυτή την ακρόαση όσον αφορά την ε, προστασία των θυμάτων που είναι βασικό σε τομέας εργασίας μου αλλά είναι και ένας πολύ βασικός τομέας πολιτικής όπου πρέπει να ενεργήσουμε ε, γρήγορα και αποτελεσματικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε και αντιδρούμε στο έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων για το είδος της κοινωνίας που θέλουμε να έχουμε και να ε, ε, δημιουργήσουμε. Είναι λοιπόν πολύ ε, σημαντικό αυτό το θέμα. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία για να δείτε λίγο το ιστορικό σε σχέση με τη μετανάστευση και την ε, διακίνηση. Φυσικά τα μεταναστευτικά φαινόμενα και γυναικών και παιδιών σχετίζονται με την διαφορετικές πραγματικότητες δεν πρέπει να δίνουμε λοιπόν απαντήσεις όχι σαν είναι ένα μόνο θέμα που ορίζεται από ένα ή δύο στοιχεία. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Δεν μπορούμε να, βάζουμε, να φτιάχνουμε πολιτικές και δράσεις που πιστεύοντας ότι υπάρχει μια ε, ομοιόμορφη απάντηση για όλες τις περιστάσεις. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι διαφορετικές οι περιστάσεις και γι' αυτό να μπορέσουμε να δώσουμε μια ταιριαστή απάντηση σε κάθε φάση. Κάποια νούμερα, τα νούμερα είναι πολύ σημαντικά και παραμένουν το μόνο αντικειμενικό ζήτημα. Δεν μπορεί κανείς να τα ερμηνεύσει όπως ε, θέλει, βοηθά αυτό στο να καταλάβουμε ποια είναι η κατάσταση πολλές φορές. Όσον αφορά το μεταναστευτικό φαινόμενο για τις γυναίκες και τα παιδιά, Βλέπουμε πως ε, σήμερα περίπου το 44,3% των μεταναστών ε, εργαζόμενων σε ολόκληρο τον κόσμο είναι γυναίκες και η αναλογία των ιδιαίτερα ε, εκπαιδευμένων ε, γυναικών ή μορφωμένων γυναικών είναι πολύ ψηλή. Η αρνητική πτυχή είναι βέβαια ότι οι γυναίκες είναι και η, πιο, η ομάδα που επηρεάζεται περισσότερο από την εμπορία. 71% ε, όλων των θυμάτων εμπορίας είναι γυναίκες. Στην Ευρώπη από τους τρία από τα τέσσερα θύματα εμπορίας είναι γυναίκες. Ε, το ποσοστό λοιπόν των γυναικών που είναι θύματα αυτού του φαινομένου είναι εξαιρετικά ψηλό παιδική μετανάστευση και αυτή αυξάνεται επίσης και ε, καθοδηγείται από διάφορους παράγοντες και εκεί έχουμε διάφορες κατηγορίες όσον αφορά τη μετανάστευση των παιδιών. Έχουμε παιδιά που μεταναστεύουν ως ανήλικοι μαζί με την οικογένεια Έχουμε παιδιά που ε, μεταναστεύουν ασυνόδευτα σε κάθε ε, ηλικία, ακόμα και πολύ πολύ μικρά παιδιά. Παιδιά που χωρίζονται από την οικογένειά τους, ε, γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειας με τους οποίους αρχικά ξεκίνησαν το ταξίδι χωρίζονται στο δρόμο, είτε γιατί κάποιος χάνεται, είτε γιατί κάποιος πεθαίνει στη διάρκεια του του, του ταξιδιού και τα παιδιά μένουν μόνα τους. Βέβαια, οι διάφορες ε, ομάδες και διάφορα είδη μετανάστευσης ε, καθορίζουν και το κατά πόσο θα εκτεθούν στην εμπορία, στην κακομεταχείριση, στην εκμετάλλευση και ένα σωρό άλλες ε, επικίνδυνες καταστάσεις. Ξέρουμε ότι το εμπόριο των ανθρώπων, ε, στοχεύει διάφορα είδη εκμετάλλευση, αλλά όσον αφορά τις γυναίκες και τα κορίτσια, το 96% των θυμάτων ε, ε, πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και μετά ένα μικρό ποσοστό για άλλους λόγους. Εκεί περιλαμβάνονται και τα ανήλικα κορίτσια ε, και γι' αυτό και είναι εξαιρετικά περίπλοκο και δύσκολο φαινόμενο. Ένα από τα στοιχεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και που θα πρέπει να απασχολήσει το Ευρωκοινοβούλιο και όλα τα κράτη-μέλη είναι ότι η εμπορία παιδιών στην Ευρώπη αυξάνεται τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Όταν μιλάμε λοιπόν για καταπολέμηση της εμπορίας και το λέμε εδώ και σε άλλες περιφέρειες της Ευρώπης κοντά ή πιο μακριά από την Ευρώπη έχουμε δίκιο αλλά είμαστε ε, προκατηλημένοι γιατί πολλά από τα προβλήματα εμπορίας συμβαίνουν εδώ στην Ευρώπη και όχι μόνο στη Βόρεια Αφρική, στα Δυτικά Βαλκάνια ή άλλες περιοχές του κόσμου κάποια στοιχεία από την μελέτη ε, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που εξετάζει την κίνηση παιδιών και νέων ε, στην Μεσόγειο και την Ανατολική Μεσόγειο που επιβεβαιώνει αυτό που είπα ότι υπάρχουν πολλαπλοί λόγοι για τη μετανάστευση και ε, επίσης το πόσο ευάλωτα είναι τα παιδιά και οι γυναίκε στο δρόμο που ακολουθούν εξαρτάται όχι μόνο από το δρόμο που θα διαλέξουν αλλά και από το αν ταξιδεύουν μόνοι του, αν ξεφεύγουν από πόλεμο, οι συγκρούσεις ή αν ε, ε, ε, αναζητούν μια καλύτερη ζωή. Υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν το επίπεδο της πιθανότητας και του, πόσο είναι ευάλωτη. και εδώ εκτίθενται περισσότερο ε, οι γυναίκες και τα παιδιά ανάλογα όπως είπαμε με το δρόμο που ακολουθούν. Βέβαια, πολλοί μετανάστες ε, που ταξιδεύουν μόνοι εκτίθεται περισσότερο στο συγκεκριμένο κίνδυνο και τα παιδιά εκτίθενται πάρα πολύ στην κατάχρηση και το εμπόριο, στην κακομεταχείριση μάλλον και το εμπόριο από εκμετάλλευση, στο εμπόριο ανθρώπινων οργάνων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. 73% των παιδιών που ταξιδεύουν ε, από την κεντρική, ε, το κεντρικό δρόμο της Μεσογείου προς την Ευρώπη έχουν αναφέρει κάποιο είδους σοβαρή κακομεταχείριση είτε σωματική είτε ψυχολογική κατά είδους, άλλου είδους. Αυτό το νούμερο θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό που γίνεται στην Κεντρική Μεσόγειο και πόσο θα πρέπει ίσως λίγο να μετακινήσουμε την προσοχή μας από το να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε με κάθε κόστος να φτάσουν οι άνθρωποι στην Ευρώπη και να αρχίσουμε να εστιαζόμαστε περισσότερο στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την ευημερία των ανθρώπων που προσπαθούν με κάθε κόστος να φτάσουν στην Ευρώπη και εκτίθεται σε τέτοιου είδους παραβιάσεις, ε, κακομεταχείριση, και να καταλάβουμε πόσο ευάλωτους τους κάνουμε όταν τους αφήνουμε να πλέουν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο πάνω σε καράβια για μέρες. Η Λιβύη είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη και ένα από τα μέρη όπου έχουμε τις περισσότερες, ε, τα περισσότερα περιστατικά κακομεταχείρισης κάθε είδους από τα παιδιά μετανάστες που είναι στην Λιβύη 70% έχουν αναφέρει ότι έχουν απαχθεί ή ότι έχουν κρατηθεί ενάντια στη βούλησή τους το 85% των παιδιών ανέφεραν ότι έχουν αυθαίρετα φυλακιστεί χωρίς ε, καμία αιτία και χωρίς πρόσβαση σε φάρμακα. Όλα τα παιδιά έχουν γίνει μάρτυρες κάποιου είδους βασανιστηρίου, δολοφονίας, σεξουαλικής ε, ε, βίας ή βίαιου εγκλήματος εναντίον των ίδιων ή εναντίον κάποιου άλλου. 63% των παιδιών που έχουν περάσει από τη Λιβύη με στόχο να μείνουν εκεί αποφάσισαν αργότερα να περάσουν προς την Ευρώπη λόγω της βίας που επικρατεί ή που υπέστησαν τα ίδια. Ως απάντηση νομίζω τρία-τέσσερα σημεία που θα πρέπει να αναφέρουμε. Πρώτον, το εμπόριο ε, ανθρώπων είναι έγκλημα, αλλά είναι και ε, προσοδοφόρα επιχείρηση. Κάποιος εμπορεύεται τους ανθρώπους, κάποιος άλλος όμως χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυτή. Και πρέπει να είμαστε το ίδιο επιθετικοί εναντίον των εμπόρων, αλλά και των διακινητών, αλλά και αυτών που συνειδητά χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των ε, διακινητών αυτών είτε είναι για εκμετάλλευση εργασίας, είτε για σεξουαλική εκμετάλλευση, είτε οτιδήποτε, θα πρέπει να διώκονται και οι χρήστες. Δεν το κάνουμε αυτό αρκετά στην Ευρώπη. Θα πρέπει να αυξήσουμε τις ενέργειές μας, θα αυξήσουμε τις έρευνες, ε, τις ποινικές διώξεις, και να επιμείνουμε με τους ιδιώτες ε, και εταίρους μας να έχουν βιώσιμες πρακτικές, επιχειρηματικές πρακτικές, δηλαδή καλύτερες συνθήκες για τους εργαζόμενους και <coughs> εργασιακή αλυσίδα χωρίς ανθρώπους που έχουν περάσει από αυτήν την αλυσίδα. Σας ευχαριστώ και δίνω τον λόγο στην κυρία ε, Βικτόρια Μιχάλκο για να μας δώσει την εικόνα ενός ανθρωπολόγου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα εστιάσω περισσότερο στην ε, εκπαίδευση για την πρόληψη. Η εμπορία ανθρώπων έχει διάφορες μορφές και η η αντιμετώπιση πρέπει να είναι εξίσου πολυδιάστατη. Η δικιά μου εργασία εστιάζεται στην Ουγγαρία και προσπαθώ να ε, δραστηριοποιηθώ στην έβρεση λύσεων για την εμπορία ανθρώπων από ανατολικά σε δυτικά. Οι νέες ε, δημοκρατίες στην Ευρώπη είναι αρκετά εύθραυστες και η... Sorry. Created during the communist... Η ομιλήτρια μιλάει πάρα πολύ γρήγορα διαβάζοντας το κείμενο, δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε. Status and no considerable economic and political position. Επιπροσθέτως, οι πληθυσμοί Ρωμά υφίστανται διακρίσεις στην Ανατολική Ευρώπη. Σε πολλές περιοχές ε, η φτώχεια επίσης ε, είναι πάρα πολύ μεγάλη στην ε, Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και την Ρουμανία συναντάμε τους στοχότερους πληθυσμούς ανθρώπων ε, στην Ευρώπη και πολλές φορές ε, θα χρειαστούν μέχρι και 7 γενιές έτσι ώστε να πλησιάσουν το μέσο εισόδημα ενώ 4,5 γενιές είναι ο μέσος όρος του ΟΣΑ. Η παράνομη μετανάστευση λοιπόν φαίνεται πως είναι η μόνη οδός και ε, ο συνδυασμός όλων αυτών δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει για το γεγονός ότι η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι τα κέντρα εμπορίας ανθρώπων. Οι αναφορές και εκθέσεις για, το, για την εμπορία ανθρώπων μας δείχνουν ανησυχητικά αποτελέσματα. Ειδικά από την νοτιοανατολική Ευρώπη βλέπουμε αυξημένες εισρωές μεταναστών οι οποίοι βρίσκουν ευκαιρία για να ε, μεταναστεύσουν στην Ευρώπη και να βρουν μια καλύτερη ζωή. Πρέπει να αντιμετωπιστούν τα αίτια του, της μετανάστευσης και να καταπολεμηθεί η ε, σύγχρονη αυτή μορφή δουλείας. Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες από διάφορους φορείς και όλοι προέρχονται ε, από, την, από το χώρο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουν τους ε, μαθητές και έχω φέρει και κάποιες πληροφορίες έντυπες οι οποίες ε, σκοπό έχουν να ενημερώσουν για αυτό που κάνουμε. Προσπαθούμε να βρούμε τις πιθανές λύσεις καταπολέμησης της σύγχρονης αυτής δουλείας αρχίζοντας από τα σχολεία μέσω της επίσημης εκπαίδευσης και διάφορων ε, μελετών. Επίσης, κάνουμε σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς ε, με σκοπό να τους ε, καταρτήσουμε ώστε να ενημερώσουν τους μαθητές τους. Πάνω από 2.000 εκπαιδευτικοί έχουν συμμετάσχει στα προγράμματά μας. Επίσης, έχουμε κάνει εργαστήρια σε πολλά σχολεία και συναντήσαμε τουλάχιστον ένα παιδί που έχει υποστεί παρενόχληση στο σχολείο ή ε, στην οικογένεια ή διάφορες άλλες μορφές εκφοβισμού. Αυτά είναι επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία που ε, δείχνουν την ευαλωτότητα των παιδιών και την αδυναμία του συστήματος να αντιδράσει. Υπάρχουν ε, πολλές περιπτώσεις κοριτσιών 13-14 ετών που πέφτουν ε, θύματα μεγαλύτερων ε, αγοριών τα οποία στη συνέχεια τις εκμεταλλεύονται σεξουαλικά. Υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό στην πρόληψη. Η πρόληψη και η ενημέρωση μπορούν να αναπτύξουν κριτική σκέψη και, έτσι, και κατόπιν αυτοπεποίθηση έτσι ώστε να ε, αποτρέπονται τέτοιες ε, και η θυματοποίηση. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ξεκινήσει αντίστοιχα προγράμματα από το 2013-2014 ε, μέσω ενημερωτικών ε, φυλαδίων, μέσω ε, ενημέρωση για το πώς να εντοπίσει κάποιο περιπτώσει εμπορίας, πώς να εντοπίζει τους διακινητές και τι να κάνει στην περίπτωση αυτή. Δεν υπάρχει κάποια, κάποιο πρωτόκολλο ακόμα ε, μόνο βέλτιστες πρακτικές. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνονται όλοι οι εταίροι και τρίτοι φορείς και τρίτες χώρες. Ε, αυτή τη στιγμή στην, ε, στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να συνεργαστούν με την Ένωση έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η εμπορία ανθρώπων. Η οργάνωσή μας επίσης ε, προωθεί την ε, συζήτηση επιγραμμικά και μη και την ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης, συνεργαζόμαστε με τις αρχές επιβολής του νόμου έτσι ώστε ε, να δραστηριοποιηθεί ε, ο νόμος για την ε, σύλληψη των ε, παραβατών αυτών. Διοργανώνουμε περίπου 12 ε, συνέδρια το χρόνο, στα οποία γίνεται ενημέρωση. Εστιάζουμε κυρίως στις πιο ευάλωτες ομάδες. Επίσης, οι μελετητές και οι πανεπιστημιακοί εστιάζουν επίσης στην ανάλυση του προφίλ των ε, διακινητών και αυτών που στρατολογούν καθώς και των πελατών τους. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε να ε, αναλάβουμε δράση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην περίπτωση όπου οι έμποροι είναι μικρές ομάδες που ανήκουν στο ίδιο κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο με τα θύματά τους. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να υπάρξει επαρκή ενημέρωση στα θύματα, προτού αυτά φύγουν από την χώρα προέλευσης. Είναι πολύ σημαντικό εκτός από τα θύματα να ενημερώνεται και ο γενικότερος πληθυσμός αλλά και οι πιθανοί αγοραστές αυτών των ε, θυμάτων. Ο, η έκθεση αυτή για την εμπορία ανθρώπων ε, συμπεραίνει ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι που συνεισφέρουν στην ε, συνέχιση της αυξητικής τάσης της εμπορίας ανθρώπων από χώρες όπως η Λιβύη, η Μολδαβία, ακόμα και η Ουγγαρία. Χρειάζεται να ληφθεί δράση σε συνεργασία με τις αρχές και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Όμως πρώτα απ' όλα χρειάζεται αλλαγή στην οτροπία και αυτό θέλει χρόνο. Χρειάζεται δικτύωση βοήθεια στις ε, χώρες από τις οποίες προέρχονται τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, ε, βοήθεια με τη μορφή μικροπιστώσεων, για παράδειγμα, και άλλων τρόπων και πάνω απ' όλα ενημέρωση. Στην αρχή σίγουρα θα χρειαστεί περισσότερο οικονομική παρά άλλου τύπου βοήθεια, όμως γίνονται βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση στόχος είναι ε, η τήρηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των ε, Ηνωμένων Εθνών και η αλλαγή στη μεταναστευτική πολιτική, η οποία πρέπει να, ε, να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Muito obrigado, ehm, Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μιχάλικο και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από πολύ κοντά τις φωνές των θυμάτων και γι' αυτό θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Εζοχέα Γκατίσε που εκπροσωπεί την ε, μη κυβερνητική οργάνωση ΙΡΟΚΟ και θα παρέμβει για 8 λεπτά. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα ότι θα μου δίνατε το λόγο αργότερα, αλλά εντάξει. Εργάζομαι για μια NGO που στηρίζει τα θύματα εμπορίας. Από την Νιγηρία αλλά και από την Ανατολική Ευρώπη. Εμείς μιλήσαμε με κάποιες γυναίκες που ήρθαν από την Μεσόγειο, περισσότερες από την Νιγηρία. Και τις ρωτήσαμε ποιο είναι το κόστος και αν ήξεραν τι κινδύνους αντιμετώπιζαν ε, μπαίνοντας σε αυτά τα σκάφη που δεν είναι ασφαλή. Και μας είπαν ότι δεν το ξέρανε ή πολλές το ξέρανε, αλλά για αυτές άξιζε τον κόπο να διασχίσουν την Μεσόγειο. Και ότι ήταν ένα θέμα επιλογής ανάμεσα στο να πεθάνουν γρήγορα στη θάλασσα ή να πεθάνουν με αργό θάνατο από φοβερή πείνα και φτώχεια. Και αυτά σας τα λέω γιατί ακριβώς η έλλειψη ευκαιριών, η βαθιά φτώχεια είναι που αναγκάζει τους ανθρώπους να φεύγουν από τις χώρες τους. Οι άνθρωποι δεν μεταναστεύουν για ένα συγκεκριμένο λόγο, δηλαδή για να σπουδάσουν, αν δεν αναγκαστούν να φύγουν από τις χώρες τους εξαιτίας συγκρούσεων, οι άνθρωποι φεύγουν επειδή οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν είναι ανυπόφορες και ψάχνουν να βρουν άλλες ευκαιρίες. Και αυτό ισχύει και για περίπου όλε τις Νιγηριανές που διασχίζουν την ε, Μεσόγειο μέσα σε τόσο επικίνδυνε συνθήκε. Οι γυναίκε λοιπόν τώρα είναι αυτές που πρώτες φεύγουν. Όντως η εμπορία ανθρώπων έχει βρει νέους ε, τρόπους να εκφραστεί οι περισσότερες γυναίκες ήδη βρίσκονται θύματα τραφικίν εμπορίας πριν καν ξεκινήσουν όταν είναι ακόμα στη Λιβύη. Λοιπόν, είπαμε ότι θέλουν να φύγουν για να βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση της οικογένειας συνήθως. Έτσι, οι γυναίκες, παιδιά, όπως ήδη γνωρίζουμε, αναλαμβάνουν αυτό το επικίνδυνο εγχείρημα. Και οι περισσότερες από αυτούς ήταν θύματα κάποιας ε, σεξουαλικής επίθεσης. Στη Σικελία, για παράδειγμα, το 2015-2016 σε καταβλισμούς έχουν ε, καταλήξει γυναίκες και μου είπαν όλες, χωρίς εξαίρεση, ήταν θύματα σεξουαλικής βίας, εκτός από άλλου είδους βίες βέβαια, έτσι. Οι περισσότερες από αυτές κατέληξαν και σε εγκυμοσύνη και οι περισσότερες είναι θέματα trafficking και έχουν καταλήξει στους δρόμους των διάφορων ευρωπαϊκών χωρών και είναι θύματα σωματεμπορίας. Λοιπόν, οι γυναίκες, τα παιδιά διασκίζουν τη Μεσόγειο, φτάνουν στους καταβλισμούς. Οι περισσότερες βρίσκονται σε επίσημους καταβλισμούς. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει με τις υπόλοιπες. Τι γίνεται με αυτές τις γυναίκες ή τα νέα κορίτσια που φτάνουν ε, με τα σκάφη αυτά και δεν είναι στους καταβλισμούς. Οι απαντήσεις που πήραμε μιλώντας με γυναίκες είναι ότι οι περισσότερες από αυτές ε, βγαίνουν από τους καταβλισμούς, κάποιος δηλαδή έρχεται, τους παίρνει από τους καταβλισμούς και τις εκμεταλλεύεται στη συνέχεια. Υπάρχουν πληροφορίες για το πώς ε, μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν στους καταβλισμούς και να τις πάρουν από εκεί. Και γίνονται θύματα λοιπόν εμπορίας, ε, είναι ήδη θύματα εμπορίας ή απλώς είναι οικονομικοί μετανάστες. Ε, διαφέρει η κατάσταση από χώρα σε χώρα. Στην Ιταλία ευτυχώ υπάρχουν προγράμματα για να στηρίξουν τα θύματα από την εμπορία αυτή ανθρώπων για να μπορέσουν να ξεφύγουν από την κατάσταση εκμετάλλευσης στην οποία βρίσκονται. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν ισχύει σε όλες τις χώρες μέλη. Και αυτό είναι το πρόβλημα πώς θα έχουμε μια ενιαία προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε τα θύματα εκμετάλλευσης και εμπορίας. Οπότε το ερώτημα που τίθεται είναι τελικά τι συστάσεις, τι λύσεις μπορούν να λειτουργήσουν. Ως μη κυβερνητικέ οργανώσεις, εμείς βλέπουμε το πράγμα ως εξής. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τι γίνεται. Είναι ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες και δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς οι αιτίες. Και ποιες είναι οι αιτίες, όπως είπα και στην αρχή, οι άνθρωποι φεύγουν από τις χώρες τους επειδή βρίσκονται σε ανυπόφορες κατάστασεις για να ζήσει κανείς και ψάχνουν να βρουν άλλες ευκαιρίες. Το ξέρουμε από τις γυναίκες που στηρίζουμε, αλλά και από τους άντρες, γιατί αν πάτε σε διάφορες Ιταλικές πόλεις, εξαιτία της άφηξης πάρα πολλών ε, μεταναστών, θα δείτε και πολλούς ε, νεαρούς άντρες οι οποίοι είναι έξω από τα μαγαζιά και ζητιανεύουν. Εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με πολλούς από αυτούς πολλά και διαφορετικά σημεία, όπως και οι συναδελφοί μου. Και τι σας λένε όλοι αυτοί, ότι αν είχαμε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε στις χώρες μας και ξέραμε ότι δεν θα βρισκόμασταν στις ίδιες καταστάσεις που μας ανάγκασαν να φύγουμε από εκεί, θα επιστρέφαμε αμέσως. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε πίσω γιατί δεν πρόκειται να βρούμε καμιά καλύτερη κατάσταση. Βέβαια το να μείνουν στην Ευρώπη επίση είναι κακό. Δεν έχουν ευκαιρίες, οι περισσότεροι δεν έχουν καν χαρτιά, οπότε τι θα γίνει. Κοιτάμε και τις κοινωνικές καταστάσεις. Δηλαδή οι ευρωπαϊκές χώρες, οι ευρωπαίοι πολίτες, πώς υποδέχονται αυτή τη ροή μεταναστών. Και βλέπουμε ένα σωρό προβλήματα τα οποία δημιουργούνται, τις κοινωνικές εντάσεις σε χώρες που δεν είχαν ποτέ μετανάστευση στο παρελθόν, τώρα ξαφνικά έχουν. Και εκεί που δεν υπήρχαν εντάσεις παλιά, τώρα υπάρχουν. Οπότε αυτό θέλουμε να δούμε και εμεί οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Η δικιά μου οργάνωση λοιπόν κάθισε και τα κοίταξε και καταλήξαμε σε κάποια προγράμματα, τα οποία είναι πιλωτικά προγράμματα, στις χώρες προέλευσης, στην Ιγυρία για παράδειγμα, από όπου προέρχονται κάποια από αυτά τα θύματα. Και ποιες είναι οι Πρώτον, όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου, σπούδασα, έμαθα για την σύμβαση ΛΟΜΕ τότε, που είχε να κάνει με τις χώρες Αφρικής, Καρεβικής και Ειρηνικού και τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόκειται για στήριξη προς αυτές τις χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναπτυχθούν περισσότερο. Λοιπόν, το αποτέλεσμα της έρευνάς μου ποιο ήταν, ότι η Σύμβαση Λομέ δεν πέτυχε αυτά για τα οποία είχε προβλεφθεί. Όχι γιατί ήταν κακιά ως αυτή καθεαυτή, αλλά γιατί δεν εφαρμόστηκε καλά. Οπότε πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο η Ευρώπη στηρίζει την ανάπτυξη στις υποανάπτυξη χώρες δεν είναι μόνο το θέμα τι κάνουν ε, οι κυβερνήσεις, είναι θέμα του τι κάνουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όταν μιλάμε για μη κυβερνητικές οργανώσεις, μιλάμε και για μη ε, κερδοσκοπικές οργανώσεις, έτσι. Όμως, αυτές οι οργανώσεις θα πρέπει να διαθέτουν πόρους για να μπορούν να κάνουν κάτι στις αναπτυσσόμενες χώρες. δεν είναι θέμα κερδοφορίας. Είναι για την κάλυψη των αναπτυξιακών προγραμμάτων ακριβώς για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Αν λοιπόν πραγματικά και ειλικρινά θέλουμε να βρούμε λύσεις στη μεταναστευτική κρίση, τότε πρέπει να επιστρέψουμε στα παλιά και να φροντίσουμε οι χώρες προέλευσης να συμμετέχουν στη βοήθεια και να είναι σε θέση οι ίδιες να βοηθήσουν τους πολίτες τους ώστε αυτοί να μην χρειάζεται να φεύγουν από εκεί. Έπειτα, τι γίνεται με τους διάφορους εθνικούς μηχανισμούς. Εδώ θα έπρεπε να υπάρξει εναρμόνιση και να υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση για τη στήριξη των θυμάτων από το τράφικινγκ. Ένα άλλο ζήτημα που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι περισσότερη στήριξη από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, την Ελλάδα για παράδειγμα και την Ιταλία. Γιατί εκεί φτάνουν πρώτα απ' όλα οι μετανάστες. Να βοηθηθούν αυτές οι χώρες λοιπόν από τις υπόλοιπες και έπειτα κοινωνικές υπηρεσίες υπάρχει αρκετή στήριξη εδώ. Είναι ένα λεπτό ζήτημα βέβαια. Δεν αντιμετωπίζεται από τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά πιστεύουμε ότι ακ... ακριβώς επειδή χρειάζεται ε, κοινωνική στήριξη για σεξουαλικά ζητήματα, γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το φροντίσουμε και αυτό αν δεν υπήρχε ζήτηση από την Ευρώπη δεν θα υπήρχαν αυτά τα θύματα σώματεμπορίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ε, τόσο εντυπωσιακή μαρτυρία αυτής της βίαιης ε, και ομής πραγματικότητα. Είναι πολύ δύσκολο, λοιπόν, πολύ σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να συνεχίσουμε όμως να το συζητάμε και να το αναλύουμε. Έχω τρεις ε, που έχουν ζητήσει το λόγο για σύντομες παρακαλώ παρεμβάσεις γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Πρώτος, η κυρία Μαϊτέ Ρουίς. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα. Καταρχά να σας πω ότι ε, σας σεβόμαστε και σας θαυμάζουμε για αυτό που κάνατε. Είμαστε σύμμαχοί σας και θέλουμε το μάξιμο των στοιχείων για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ακριβώς ε, τι συμβαίνει. Θα θέλαμε να ξέρουμε αν έχετε αριθμητικά στοιχεία. Εκτιμήσεις. Πόσες χιλιάδες παιδιά και γυναίκες έχουν ε, επηρεαστεί από αυτά που μας είπατε στην, στην περίπτωση των παιδιών που που πέφτουν θύματα εμπορίου ανθρωπίνων οργάνων, έχετε στοιχεία. Γιατί για μας, για να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη, θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στοιχεία. Γιατί η, πρέπει η κοινή μας γνώμη να αποκτήσει και πάλι ανθρωπιά να ε, μπορέσει να δει τι πραγματικά συμβαίνει, ε, να συγκινηθεί. Και έπειτα γίνεται λόγος για 9.000 ε, κόσμο που έχει έρθει από την Μεσόγειο. Είναι περισσότεροι. Ξέρετε εσείς αν είναι περισσότεροι οι γυναίκες και τα παιδιά πόσα παιδιά είναι αυτά που έχουν επηρεαστεί για να στείλουμε ένα πολύ πιο έντονο μήνυμα για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο ανθρώπινη την ε, μάτια έπειτα. Ποιο συμβαίνουν ε, πράγματα τα τελευταία τρία χρόνια. Στην Κατάνια πριν από λίγες μέρες μας έλεγαν ότι είχε μειωθεί ε, πάρα πολύ ο αριθμός των αφήξεων από την Λιβύη, ότι έρχονται περισσότεροι από την, ε, την Ισία. Ξέρουμε ότι στη Λιβύη κρατούνται τα παιδιά, οι άντρες, οι γυναίκες, όλοι. Μπορείτε να μας πείτε τι συμβαίνει. Σας ευχαριστώ και πάλι ε, και συγχαρητήρια για το έργο σας. Ευχαριστούμε. Λόπες Ακυγιάρ. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση για τον κύριο Αμπρόζη. Αυτή στις συνεδριάσεις είναι ε, ε, συναρπαστικές. Κάποιες φορές ε, φτιάχνουμε, νομοθετούμε, κάποιες φορές τσακωνόμαστε για καυτά ζητήματα και κάποιες φορές ακούμε από πυρεγνώμονες μάρτυρες που πρέπει να προσέξουμε. Ακούμε μόνο και μας δίνεται τροφή προσκέψη. Και αυτό συμβαίνει όταν πρόκειται για το εμπόριο ανθρώπων και την πετάλευση ανθρωπίνων όντων και ακριβώς το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι ακριβώς αυτό που είπατε ότι όταν μιλάμε για την εκμετάλλευση των γυναικών σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών έχουμε την τάση να είμαστε κάπως μετριοπαθείς και να σκεφτόμαστε ότι ναι, κάπου αλλού όμως γίνονται όλα αυτά. Λιβύη εκμεταλλεύεται τις γυναίκες για σεξουαλικούς σκοπούς, αλλά αυτό συμβαίνει εδώ, στην άλλη όχθη, την ευρωπαϊκή όχθη της ε, Μεσογείου, συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη και κάτι πρέπει να γίνει. Και σύντομα θα ήθελα να τονίσω μια δική μου εμπειρία. Βρισκόμουν, που ήμουν κάποτε υπουργό ε, Δικαιοσύνης ε, του Βασιλείου της Ισπανίας, κράτος μέλος και ήμουν μέλος του Συμβουλίου των Υπουργών που ε, ασχολήθηκε με την ποινικοποίηση της πορνείας σε ολόκληρη την Ένωση. Υπήρχε ένα κράτος μέλος που τόνισε την ιδέα η Σουηδία και υπήρξε μια έντονη ε, συζήτηση ε, για την ε, πιθανότητα δίωξης με το, μέσω του ποινικού δικαίου δίωξης της πορνείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι, είναι δύσκολο όσον αφορά την, το ποινικό δίκαιο και την πολιτική την, που θα σκεφτεί κατά του εγκλήματος. Όμως όσον αφορά ε, το γεγονός ότι η κατάσταση έχει μόνο επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι ε, μεγάλη επιχείρηση η πορνεία. Σε κάποια κράτη μέλη εκμετάλλευση των γυναικών για εγκληματικού λόγους, για την πορνεία δηλαδή, έχει γίνει σε ορισμένες χώρες το νούμερο, ε, το, η νούμερο ένα προσοδοφόρα εγκληματική ε, επιχείρηση. Είναι ε, μαζί με διάφορες άλλες ε, δραστηριότητες. Αυτή, αυτό είναι που απασχολεί το οργανωμένο έγκλημα. Εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί τώρα υπάρχει νομική βάση, πράγμα που δεν υπήρχε πριν από 10 χρόνια, πριν αρχίσει να ισχύει η Λισαβόνα. Δεν ίσχυε το 2004 όταν εγώ ήμουν Υπουργός Δικαιοσύνης. Τώρα όμως έχουμε νομική βάση για την ποινικοποίηση των σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων με την νομοθέτηση ποινικού δικαίου και την άσκηση ποινικής ε, πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ παρακαλώ να είστε πιο σύντομοι στη διατύπωση των ερωτημάτων σας για να μπορέσουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις των ε, προσκεκλημένων μας. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ το τον συνάδελφο που έθιξε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και σας ευχαριστώ επίσης που μιλάτε για το θέμα της ζήτησης. Είμαι... Ε, ήμουν ε, μέρος, ε, συμμετείχα μάλλον στη διατύπωση αυτής της νομοθεσίας και θα ήθελα όντως να τιμωρηθούν αυτοί που αγοράζουν την υπηρεσία ε, του εμπορίου. Δεν μπορέσαμε τότε να το περάσουμε. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε στο μέλλον. Είμαι σε επαφή με διάφορες ε, θελοντικές οργανώσεις και έχω συμμετάσχει σε, ε, στις περιπολίες της αστυνομία. Έχουμε συναντήσει πολλές ε, πόρνες από την Ναγυρία και μάλιστα έχω και επαφές με μια οργάνωση που ονομάζεται Ταλίτα. είναι εθελοντές και ασχολούνται με τα θύματα της σωματεμπορίας στην Σουηδία. Χρειάζεται ένα δίκτυο των ΜΚΟ, χρειάζεται να έχετε τη δύναμη να αντιδράσετε, να θέσετε, να, να δώσετε τα καλά παραδείγματα. Νομίζω λοιπόν πως είναι πολύ σημαντικό οι οργανώσεις στην Ένωση που ασχολούνται με αυτά τα θέματα να δικτυωθούν μεταξύ τους. Ίσως να ήδη να έχετε επαφές, δεν ξέρω, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να έχετε ε, καλά δίκτυα και να είστε δικτυωμένοι με οργανώσεις στην ε, Νιγηρία, στη Λιβύη επίσης, γιατί ξέρουμε πως τα θύματα του εμπορίου συχνά επιστρέφουν και θα θέλαμε να είμαστε βέβαιοι ότι επιστρέφουν υπό καλές συνθήκες. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Έχω μία ερώτηση ε, για την κυρία Ιρόκο. Αυτή είναι Ιρόκο. Δεν τη λένε Ιρόκο. Είναι εκ μέρους της ε, οργάνωσης Ιρόκο. Υπάρχει, υπάρχουν μεγάλες ροές ε, προς τη Δύση. Στην Πολωνία επευλήθη ε, μία μορφή ε, αυστηρής νομοθεσίας, η οικονομία ε, είχε προβλήματα. Στη χώρα υπήρχε μεγάλη ισροή μεταναστών από χώρες στις οποίες είχε επιβληθεί στρατιωτικός νόμος. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά προβλήματα, αλλά Εμένα θα με ενδιαφέρει πιο πολύ να μάθω για τους λόγους για τους οποίους φεύγει ο κόσμος και γιατί φεύγει ο κόσμος από την Νιγηρία. Γιατί υπάρχει τέτοια μεγάλη εισρωή ανθρώπων από την Νιγηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νιγηρία είναι μια πλούσια χώρα, έχει πρώτες ύλες και αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Επίσης, Αναφερθήκατε στο γεγονός ότι τα θύματα είναι συνήθως γυναίκες οι οποίες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες τους. Πώς αρχίζει όμως η όλη μετακίνηση, πώς ξεκινά. Και άλλη μια ερώτηση. Σε ποιους άλλους προορισμούς ε, πηγαίνουν οι ε, μετανάστες από την Ιγυρία. Έχουν οικογένειες που ήδη μένουν στην Ευρώπη. Η Πολωνία έχει σχέσεις με την Ιγυρία. Για παράδειγμα, ένας ε, ποδοσφαιριστής εθνικής ομάδας Πολωνία κατάγεται από την Ιγυρία και ένας ε, συνάδελφός μου στο Κοινοβούλιο της Πολωνίας ε, είναι από την Ιγυρία. Έχουμε λοιπόν δεσμούς με τη χώρα αυτή. Θα ήθελα όμως να επαναλάβω την ερώτηση μου. Ποιοι είναι οι λόγοι της μετανάστευσης από την Ιγυρία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπιόρκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τους προσκεκλημένους και τους εμπειρογνώμονες. Το θέμα αυτό απασχολεί την Επιτροπή Ισότητας εδώ και πολύ καιρό και μας εμπνέει η δουλειά που κάνετε, όχι μόνο εσείς που είστε εμπειρογνώμονες, αλλά και οι ε, εθελοντικές οργανώσεις. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να αποκαταστήσουμε ε, την προσοχή του κοινού στα θέματα αυτά. Όποιος έχει πάει σε, στρατόπεδα υποδοχής ε, θα έχει παρατηρήσει τι συμβαίνει εκεί. Υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι είναι κλειδωμένοι εκεί και περιμένουν να πελαθούν. Και για μένα είναι σαφές ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι θύματα εμπορίας. Και αντί να λαμβάνουν τις υπηρεσίες τις οποίες δικαιούνται, ε, Του κλείδαν παρόν σε αυτά τα στρατόπεδα και είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα και είναι πολύ σημαντικός αυτός ο μηχανισμός μεταρρύθμισης έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και να μην ε, φυλακίζονται. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε περισσότερο τις εθελοντικές οργανώσεις και οργανώσεις όπως την είπατε του ΕΕ, τους πρόσφυγες και να στηρίξουμε επίσης τα σημεία ε, άφηξης όπου και ε, λαμβάνει η χώρα η εμπορία ανθρώπων σε μεγαλύτερο ποσοστό. Επίσης πρέπει να δούμε και τις λύσεις μακροπρόθεσμα. Έχουμε συζητήσει στο παρελθόν ε, για το ότι θέλουμε διάφορες μορφές συνεργασίας με ε, χώρες, ε, τρίτες χώρες, όπως χώρες της Αφρικής και χρειάζεται λοιπόν να διαθέσουμε και κονδύλια όχι μόνο στην καταπολέμηση αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών αυτών και πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την μετανάστευση. Αυτή τη στιγμή η Εκεί ε, δεν χαρακτηρίζεται από ευνοϊκό κλίμα για αυτό το θέμα. Είναι τρομερό το ότι υπάρχουν τόσες νόμιμες οδοί, μετανα... δεν υπάρχουν νόμιμες οδοί μετανάστευσης ε, και αυτό είναι λυπηρό. Στη Σουηδία, τη χώρα μου, υπάρχουν μέτρα τα οποία ήταν αρκετά αποτελεσματικά ε, όσον αφορά την πρόληψη της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών, γιατί εμείς εστιάζουμε στη ζήτηση και δεν ποινικοποιούμε ανθρώπους οι οποίοι ε, εκτίθενται στην πορνεία. Γι' αυτό λοιπόν και τα αποτελέσματά μας είναι καλά. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να ρωτήσω ποιοι ε, είναι οι κυριότεροι προορισμοί των ε, θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και ποιες είναι οι χώρες προέλευσης ε, των θυμάτων αυτών. Κοιτάξτε, πρέπει δυστυχώς να ζητήσω από τους ομιλητές να είναι, πιο σύντομοι γιατί ε, ε, δεν θα μπορέσουν να δώσουν τις απαντήσεις τους διαφορετικά και να ακούσουμε και τη δεύτερη συνεδρία. Παρακαλώ πάρα πολύ λοιπόν σε δύο λεπτά να δώσετε την απάντησή σας ε, όσο γίνεται πιο σύντομα. Σας ευχαριστώ. Πολύ σύντομα θα προσπαθήσω να απαντήσω. Το θέμα των γυναικών και πώς φεύγουν. Συνήθως κάποιος τις πλησιάζει, που δεν είναι από τους λαθροδιακινητές, έτσι στην Νιγηρία την ίδια. Βέβαια η κυβέρνηση έχει φτιάξει μια task force ήδη από πέρυσι από τον Αύγουστο που προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και να εντοπίσει τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι μπορεί να μην είναι ε, λαθροδιακινητές αλλά αυτοί είναι οι οποίοι πιέζουν, είναι αυτοί που πηγαίνουν επίσης στη Λιβύη το Φεβρουάριο από όσο ξέρω κάπου 7.000 επέστρεψαν το θέμα λοιπόν πάντα είναι θέμα πόρων. Δηλαδή πώς οι άνθρωποι αυτοί που έχουν φτάσει στην ε, Λιβύη, πώς θα επιστρέψουν πίσω στην Ιγυρία. Τώρα, για τις οικογένειες που ήδη βρίσκονται στην Ευρώπη, είναι πάρα πολύ λίγες. Δηλαδή, οι άνθρωποι που περνάνε από τη Μεσόγειο δεν έχουν συνήθως οικογένειες. Αυτοί που έχουν οικογένειες δεν περνάνε από τη Μεσόγειο με τέτοιο επικίνδυνο τρόπο, ακολουθούν άλλες νόμιμες οδούς για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Ναι, το ξέρω ότι η Πολωνία έχει δεσμούς με την Ιγυρία. Και ακριβώς γι' αυτό θα μπορούσε η Πολωνία να στηρίξει περισσότερο την Νιγηρία στις προσπάθειές της, ώστε να σταματήσει αυτή η λαθροδιακίνηση. Το θέμα τώρα της ροής και γιατί υπάρχει τέτοια μετανάστευση δεδομένου ότι η Νιγηρία είναι πλούσια χώρα. Ναι, τεχνικά όντω είναι πλούσια χώρα η Νιγηρία, αλλά το ξέρουμε και εγώ από την Νιγηρία είμαι. Γνωρίζουμε πολύ καλά τους λόγους για τους οποίους ο πλούτος της Νιγηρίας δεν έχει οδηγήσει σε ανάπτυξη, σε καλή κατάσταση στη χώρα. Είναι διαφθορά και όλοι το ξέρουμε. Νομίζω ότι μπορούμε ανοιχτά να το παραδεχτούμε αυτό. Και υπάρχει επίσης και η ευρωπαϊκή προσέγγιση θα έπρεπε η Ευρώπη να ζητήσει από την Ιγυρία να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Έπειτα, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και οι πόροι του. Εμεί, όπω είπε και η Σουηδή Ευρωβουλευτής, δεν έχουμε αρκετούς πόρους ως μη κυβερνητικέ οργανώσει για να εκτελέσουμε το έργο μας και αυτό μας εμποδίζει. Τώρα χώρες που πάνε περισσότεροι μετανάστες είναι Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, Αυστρία. Εκεί κυρίως καταλήγουν. Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Ελβετία. Είναι εύκολο να αγοράσει κανείς γυναίκες για σεξ. Εξού και εκεί φτάνουν τα περισσότερα θύματα. Εκεί που υπάρχει αλλαγή στην νομοθεσία, εκεί υπάρχει και μεγάλη μείωση των αφήξεων. Από πού? Από αραβικές χώρες. Και εκεί πολλές γυναίκες εκμεταλλεύονται σεξουαλικά. Αυτά, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μιχάλκο, σύντομο σχόλιο. Ευχαριστώ. Ναι, θέλω να αφήσω χρόνο και στους άλλους. Οπότε θα απαντήσω μόνο στην τελευταία ερώτηση για την εκπαίδευση, τη μόρφωση. Επειδή μίλησα εγώ γι' αυτό. Η ανάπτυξη, πιστεύω, και η αντιμετώπιση των αιτιών της μετανάστευσης είναι το πιο σημαντικό. Έτσι θα μειωθεί η σύγχρονη αυτή δουλεία που συνδέεται με την μετανάστευση. Από την άλλη, στην Ευρώπη δεν θα έπρεπε να, να δούμε τη μετανάστευση μόνο σαν πρόβλημα ασφάλειας. Θα έπρεπε να δούμε πώς μπορούμε να φροντίσουμε για νόμιμες οδούς μετανάστευσης, νόμιμους τρόπους. Τη στιγμή που υπάρχει περιθώριο για εργασία για ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να έρθουν από την Αφρική, από την Ασία ή απαλού για να βρούνε δουλειά στην Ευρώπη. Πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε ότι η μετανάστευση αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο εν μέρη τουλάχιστον, και άρα πρέπει να δημιουργηθεί ο κατάλληλο χώρο για νόμιμη μετανάστευση. Ευχαριστώ, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε κύριο Σαμπρόζη. Ευχαριστώ και εγώ. Πολύ σύντομα θέλω να αναφερθώ στα στοιχεία και τα νούμερα. Εννοείται, εντάξει, ευχαρίστω. Σα έδωσα ήδη μερικά. Ναι, έχουμε στοιχεία, αυτά που ζητήσατε δηλαδή και μπορώ να τα δώσω στον πρόεδρο της Επιτροπής σας άμα θέλετε και μπορεί να τα διανύμει και στα μέλη εφόσον σας ενδιαφέρουν. 35.000 περίπου παιδιά είχαμε πέρυσι, για παράδειγμα, 23% αυτών πριν φτάσουν στην Ευρώπη ήταν ήδη θύματα Κάποιον... Ε, βίων φαινομένων. Αυτά τώρα για τις αφήξεις από τη Βόρεια Αφρική που λέτε ότι έχουν μειωθεί οι αφήξεις. Αυτό ίσως είναι το καλό. Το κακό όμως, μάλλον τα κακά ναι, είναι δύο. Πρώτον, αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται κάπου αλλού, στη Βόρεια Αφρική, είτε στη Λιβύη, είτε αλλού και θα έπρεπε να μας ε, απασχολήσει αυτό γιατί οι συνθήκες τις οποίες ζουν εκεί όπου βρίσκονται στη Βόρεια Αφρική δεν είναι καλές και άρα δεν θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει μόνο ο αριθμός αφήξεων, θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει και η κατάσταση στην οποία ζουν αυτοί οι οποίοι δεν φτάνουν σε μας. Και το άλλο κακό είναι ότι παρά την μείωση των αφήξεων στην Ευρώπη, το ποσοστό θανάτων σε σχέση με τις αφήξει έχει αυξηθεί, έχει διπλασιαστεί στην πραγματικότητα. Δηλαδή, λιγότεροι άνθρωποι φτάνουν, περισσότεροι άνθρωποι σε ποσοστό χάνουν τη ζωή τους. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό. Δεν είναι δυνατόν από το 2000 στη Μεσόγειο έχουν χαθεί πάνω από 40.000 άνθρωποι. Αυτά τα νούμερα θυμίζουν πόλεμο, έτσι και είναι στις πόρτες μας, δίπλα μας. Αυτή είναι μια ανησυχία που πρέπει να μας απασχολήσει όλο και περισσότερο. Και ναι, είμαστε πεπισμένοι και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πεπισμένη για το ότι όντως πρέπει να υπάρξει περισσότερη ποινικοποίηση και δίωξη όλων αυτών οι οποίοι χρησιμοποιούν επίτηδες είτε την πορνεία είτε την παράνομη εργασία στη Γεωργία, ας πούμε, στην Νότιο Ιταλία, είτε αλλού, γιατί το βασικό είναι ότι πρόκειται για business. Και ο μόνος τρόπος να σταματήσει αυτή η επιχειρηματική εντό εγωγών δραστηριότητα είναι να μην υπάρχει ζήτηση. Όσο υπάρχει αγορά και ζήτηση, προφανώς και θα υπάρχει αυτό. Κάποιοι θα προσπαθούν να βγάλουν χρήματα από αυτό. Άρα πρέπει να διώξουμε τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών. Και αν οι άνθρωποι που φτάνουν σε εμά θέλουν ένα μέλλον και δέχονται να τύχουν εκμετάλλευση μέχρι ένα σημείο, έτσι καλώ είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν το λαθροδιακίνητη, Γιατί αλλιώ πώ θα φτάσουν στην Ευρώπη να βρουν δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην ε, Ευρώπη την εποχή των Ναζί, οποιοδήποτε ήθελε να γλιτώσει, ε, πώ θα γλίτωνε, θα έφευγε με κάποιο παράνομο τρόπο για να γλιτώσει. Άρα είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Και δυστυχώ σε τέτοια κατάσταση βρίσκονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Αν λοιπόν δεν ε, κάνουμε αυτά που σα είπα, δεν θα ξεφύγουμε από το πρόβλημα. Τώρα, δηλαδή, τα χρήματα που πάνε για την ασφάλεια, άμυνα κτλ. Τώρα δεν ξέρω αν είμαι αφελή ή ιδεαλιστή. Πάντω είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι η καλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε στην ασφάλεια δεν είναι οι φράχτες και οι φυλακές, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα να εφαρμόζονται παντού όπου παραβιάζονται ανά τον κόσμο. Και αυτά λέει και η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εξάλλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά προβλέπει. Και ο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί έναν από του πυλώνε πάνω στου οποίου έχει χτιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε, αν θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Όσο ασχολούμαστε μόνο με το τελευταίο κομμάτι του φαινομένου, τότε θα γυρνάμε γύρω-γύρω και το πρόβλημα θα παραμένει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ τους τρεις ε, που ε, πήρατε το λόγο και περνάμε στο επόμενο, στην επόμενο πάνελ να αλλάξουν οι ομιλητές. Παρακαλώ τους επόμενους ομιλητές να έρθουν ε, και να ανεβούν εδώ. Κυρία Σινόβα. Ε, ε, ε, η κυρία Βασιλιάδου και η κυρία Γιαρμπουσινόβα. Estando a mesa já eh, instalada, estaríamos em condições de prosseguir para o segundo eh, painel. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε με αυτό το καινούριο πάνελ που αφορά τα πιο συγκεκριμένα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν κατά του ε, εμπορίου ανθρώπων. Δώσω λοιπόν ήδη το λόγο στην κυρία Μύρια Βασιλιάδου που είναι συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον, ε, στις προσπάθειες που γίνονται εναντίον της ε, εμπορίας ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις δύο επιτροπές ε, που συνεδριάζουν σήμερα για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνουν για τον τομέα αυτών. Σήμερα εστιάζουμε στην εμπορία γυναικών και παιδιών στα πλαίσια, στο πλαίσιο της μετανάστευσης, που είναι η νέα μορφή δουλείας της εποχής μας. Ε, θα ήθελα να δω, διακάνω κάποιους ε, διαχωρισμούς σε θεματικές Πρώτα, εμπορία γυναικών και παιδιών. Γνωρίζουμε από στατιστικά στοιχεία της ε, Eurostat και της Ευρωπολ ότι τα δύο τρίτα των θυμάτων εμπορίας είναι γυναίκες και κορίτσια. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνούμε. Επίσης, γνωρίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών και των κοριτσιών, αν όχι όλες, ταξιδεύουν στην Ευρώπη για σκοπό σεξουαλική εκμετάλλευση. εκμετάλλευσης. Είναι κάτι που δεν μας βολεύει να λέμε, αλλά είναι η αλήθεια. Δεδομένη τη σημασία που έχουν τα στατιστικά στοιχεία, να πω ότι παρατηρείται 60% αύξηση στην εμπορία γυναικών από την Νιγηρία ε, στην Ιταλία μέσω της Λιβύης. Ε, από το 2014 μέχρι τώρα, λοιπόν, 60% ε, αύξηση ε, της εμπορίας γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση. Είναι Πολύ ξεκάθαρα λοιπόν αυτά τα στοιχεία. Αυτό όμως που παραμένει ε, ασαφές είναι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας. Ακούσαμε σήμερα το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ε, τα ίδια λόγα, λόγια με αυτά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπάθησαν να ανταποκριθούν στο θέμα αυτό, στο πρόβλημα αυτό, ε, εστιάζοντας βέβαια περισσότερο στα παιδιά παρά στις γυναίκες. Ε, για να δανειστώ και εγώ μερικά από τα λόγια του Προέδρου. αλήθεια, τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Ε, έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλά συνέδρια και εκδηλώσεις για το θέμα αυτό. Υπήρξα υπεύθυνη για χρηματοδότηση αρκετών φορέων από μη κυβερνητικέ οργανώσεις μέχρι διεθνείς οργανισμούς ε, που ασχολούνται, στον, ε, που δεστηριοποιούνται στο χώρο αυτό. Και τα τελευταία ε, χρόνια έχω συμμετάσχει σε άπειρα συνέδρια. Όμως, πόσα από όλα αυτά τα συνέδρια, πόσες από όλε αυτές τις δράσεις λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου. Πόσα από ε, πώς από αυτές τις αποφάσεις λοιπόν έχουν υπόψη τη, τα αριθμητικά αυτά στοιχεία. Ίσως οι συνάδελφοι να έχουν μια απάντηση σε αυτό. Ε, επίσης μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μια, μια μορφή ε, εγκλήματος ε, αρκετά αξιόπινης πράξης και ταυτόχρονα σεξουαλική εκμετάλλευση. Υπάρχει εξαιρετική νομοθεσία από το 2011 ο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει μία έκθεση μεταφορά ε, το, σε νομοθεσία στο Εθνικό Δίκαιο και σήμερα ε, είμαι εδώ. Να σας πω τον περασμένο Ιανουάριο ε, ήμουν πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ε, μιλήσω εκείνη τη φορά για τις ε, παραβιάσεις ε, του, της νομοθεσίας. Ε, πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ροή του χρήματος τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά της Ένωσης. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένες δράσεις για ε, το θέμα αυτό, διότι είναι η τελευταία ε, οργάνωση που προσπαθεί να ασχοληθεί, που ενσκύπτει στο πρόβλημα των γυναικών των κοριτσιών και των αγοριών, γιατί υπάρχει σαφής διαχωρισμό. δεν μιλάμε για παιδιά, αλλά για κορίτσια και για αγόρια εδώ. Έχει διαφορά. Το Ινστιτούτο Ισότητας Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται εδώ και πολύ καιρό με το πώ ε, θα μεταφερθεί η σχετική οδηγία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πώ θα προστατευτούν τα ευάλωτα παιδιά από τις διαδικασίες αυτές και ε, την περασμένη εβδομάδα οδηγηθήκαμε στην υπογραφή μιας κοινή δήλωσης από 10 ευρωπαϊκούς οργανισμούς που ε, στόχο έχουν την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων. Αυτό συμπεριλήφθηκε σε μια ανακοίνωση της Επιτροπής και μας χαροποιεί ιδιαίτερα διότι υπάρχει αγαστή συνεργασία, δικαστική ε, συνεργασία μεταξύ των ε, αρχών, επιβολής του νόμου και όλων των κοινωνικών φορέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης πρόσφατα ξεκίνησε μία πρωτοβουλία σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη για να αντιμετωπίσει την βία κατά των γυναικών. Και ένα από τους τομείς εστίασης είναι η εμπορία ανθρώπων. Η Κομισιόν φαίνεται πως αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος ε, παγκόσμιος ε, ε, φορέας ο οποίος ασχολείται συστηματικά με το ζήτημα της διάστασης του φύλου στο, στην ε, περίπτωση της εμπορίας ανθρώπων. Μετά, χρηματοδοτούμε ε, διάφορες δράσεις κατά της εκμετάλλευσης ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι διπλασίασε τη χρηματοδότηση για τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η εμπορία ανθρώπων ε, φυσικά έχει διάφορες διαστάσεις. Σεξουαλική εκμετάλλευση, εμπόριο οργάνων, ε, εκμετάλλευση για εγκληματικές δραστηριότητες, ε, δουλεία κτλ. Φυσικά όμως υπάρχουν ορισμένοι ιδιαίτερα σχετικοί τομείς και να περάσω τώρα στον δεύτερο άξονα της ομιλίας μου με θέμα τη μετανάστευση. Η μετανάστευση είναι κάτι που προκαλεί ε, έντονες ανησυχίες παγκοσμίως. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εμπορία ανθρώπων στην Ευρώπη ε, αφο... ότι τα δύο τρίτα μάλλον των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ε, είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ε, πρέπει να εθελοτυφλούμε άλλο. Ούτε ε, πρέπει να αρκούμαστε στο να λέμε ότι υπάρχει μία τάση να χρησιμοποιούμε ορολογία για να καλύπτουμε την ουσία. Μετά, ε, να μιλήσω τώρα για την νέα μορφή δουλείας. Λυπάμαι που το λέω καταρχάς, αλλά δεν υπάρχει κάποια νέα μορφή δουλείας. Όταν μιλάμε για ευάλωτους μετανάστες, τι ακριβώ εννοούμε. Δεν υπάρχουν ευάλωτοι μετανάστες. Ποια είναι η νέα μορφή δουλεία και ποια ήταν η παλιά. Ε, υπάρχει νέα μόδα και παλιά μόδα. Καλύτερα να κρατήσουμε τη, τους νομικούς ορισμούς ε, που έχουν δρεωθεί διεθνώς. Και να μην ξεχνάμε, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές και τους ευχαριστώ γι' αυτό, ότι το θέμα ε, είναι απλό. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιο είναι ευάλωτο πρέπει να τον εκμεταλλευόμαστε. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε δεδομένο ότι εντάξει, το κορίτσι αυτό 10 χρονών στην, από την Ιγυρία ήταν στο δρόμο, είναι ευάλωτο, τι να κάνει κανεί. Όχι. Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο θα λύσουμε τα προβλήματα δεν είναι δικαιολογία το ότι επειδή κάποιος είναι φτωχό, επειδή έχει περάσει βίο παρελθόν, επειδή προέρχεται από μέρη όπου υπάρχουν διενέξει περιβαλλοντικές καταστροφές, ε, ο, αναμένεται να πέσει θύμα εκμετάλλευση. Καλύτερα να αντιστρέψουμε λοιπόν ε, τα πράγματα και ε, ακούστε εδώ τι έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Η ευαλωτότητα, ο βάλατος χαρακτηρά δεν είναι η αιτία της εμπορίας. Όπως είπε και η συνάδελφος από την Ιγυρία, ο κόσμος μεταναστεύει για διάφορους λόγους. Όμως, όσο κάποιος εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους, όσο κάποιος εκμεταλλεύεται σεξουαλικά, δηλαδή αυτό είναι ένας ωραίος να πούμε βία σε ένα κορίτσι για πέντε ευρώ στο δρόμο, όσο ε, υπάρχει εκμετάλλευση, εκμεταλλευτές και ε, πελάτες ε, των εκμεταλλευτών αυτών, δεν θα αλλάξει τίποτα. Οι συνάδελφοι της Ευρωπόλ μας ε, λένε πως ε, το κέρδος από την εμπορία ανθρώπων ε, ανέρχεται σε 30 δισεκατομμύρια. Όσο λοιπόν συνεχίζουν αυτές οι πρακτικές δεν πρόκειται να σταματήσει και να αλλάξει τίποτα. Πρέπει να ακολουθήσουμε τη ροή του χρήματος, να σταματήσει η ατιμορρησία επιτέλους και να απαιτήσουμε από τα κράτη-μέλη τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει τίποτα να ποινικοποιήσουν έστω εκείνους όσοι χρησιμοποιούν εν γνώση τους τους καρπούς του εγκλήματος. Δεν πρέπει να ποινικοποιούνται ε, οι λάθος άνθρωποι, αλλά εκείνοι που ε, εθελοντικά χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του εγκλήματος. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ε, φυσικά και ε, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν κυρώσεις. Αν πάρεις ας πούμε μία ε, τσάντα παράνομα από κάποιον πλανόδιο πολιτή θα ε, τιμωρηθεί ποιος αυτός που πουλά τα παράνομα προϊόντα. Έχουμε έναν αριθμό 9.000 γυναικών και κοριτσιών από την Ιγυρία που εκτιμάται ότι έχουν πέσει θύματα εμπορίας σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Ε, ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια ευρώ έχουν κερδίσει οι διακινητές τους, οι σωματέμποροι. Μπορείτε να κάνετε μερικές απλές μαθηματικές πράξεις για να βρείτε πόσοι εποφελούνται από αυτές τις εγκληματικέ ενέργειες και πόσοι τιμωρούνται. Και αν σα είναι δύσκολο να σας πω ότι κανείς δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Βασιλιάδου. Να δώσω τώρα το λόγο στην Μαρίνα Γιαρμπουσινόβα που είναι ειδική εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ και συντονίστρια για την καταπολέμηση του εμπορίου των ανθρώπων Παρακαλώ να ε, περιοριστείτε στα 8 λεπτά ώστε να μας μείνει χρόνος για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι τιμή μου που σήμερα ε, μίλησα για αυτό ναι, με καλέσατε για να μιλήσω για αυτό το θέμα και θέλω να επενέσω την Επιτροπή Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών καθώς και την Επιτροπή Γυναικών και Ισότητας που διατηρούν την έμφαση σε αυτό το θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό. Όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές, το εμπόριο ανθρώπων συνεχίζει να αυξάνεται και διαπιστώνουμε πως ε, συμβαίνει σε διάφορα σενάρια. Καταρχάς, ε, ε, αναγκασμένοι να κινηθούν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν, εκτίθενται σε λίτρα, σε απαγωγές, σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Φτάνοντας στην Ευρώπη, όμως, το εμπόριο συνεχίζεται. Δεν περιορίζεται μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε όλα τα κράτη και στο, στα κράτη του ΟΑΣΕ και αυτό λόγω της ευάλωτης κατάστασης ε, στην οποία βρίσκονται οι μετανάστες. Επίσης, αυτοί που είναι οι τυχεροί και φτάνουν στην Ευρώπη και ενώ περιμένουν ε, την ε, διεκπαιρέωση της αίτησής τους, είτε αυτοί οι οποίοι ε, γλιτώνουν από πνιγμό, ήδη είναι ευάλωτοι και φυσικά πολλοί εξ αυτών κινδυνεύουν να πέσουν ε, στη πλοκάμια των ε, ανθρώπων που τους εκμεταλλεύονται και στα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος και να γίνουν θύματα σεξουαλικής βίας και κακομεταχείρισης. Φυσικά όλα αυτά τα σενάρια χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες από τις εθνικές αρχές, από την κοινωνία των πολιτών και από τη διεθνή κοινότητα. Και το θέμα που συζητάμε σήμερα και συζητήθηκε και πριν δύο μέρες στο πλαίσιο της ε, Επιτροπής ε, του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΑΣΕ και του ΟΗΕ. Συχνά, όπως είπατε και εσείς, αποτελεί δυστυχώς τακτικό θέμα συζήτησης. Δυστυχώς όμως, παρά από την καλή, την καλή νομοθεσία που ισχύει σε πολλά κράτη, ανεξάρτητα από τη δέσμευση που διεθνώς έχει εκφραστεί, η ε, εμπορία παραμένει απειλή για την ανθρώπινη φυλή. Και η εφαρμογή των νομοθεσιών θα πρέπει να γίνεται καλύτερα. Και αυτό πάντοτε το λέω στις επισκέψεις μου στις χώρες γιατί μιλάμε φυσικά για μέτρα κάνουμε πολύ μεγάλη δουλειά με τα 57 κράτη για να επιμείνουμε στην καλύτερη εφαρμογή, στην καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας και να βοηθήσουμε τα κράτη να βοηθήσουν, να, να βελτιώσουν τον εντοπισμό των θυμάτων της ε, εμπορίας. Είναι πρόβλημα σε όλα τα κράτη γιατί αν και οι διεθνείς οργανισμοί ΑΕΛΟ, IOM μιλούν για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πέφτουν θύματα εμπορίας ή τα στατιστικά στοιχεία που λαμβάνουμε από τις χώρες μέλη μας είναι πολύ χαμηλά. Και πολύ χαμηλός είναι και ο αριθμός των ε, εντοπισμένων και ε, υποδίωξη διακινητών. Θα πρέπει λοιπόν να αυξηθεί και η ανταπόκριση της ποινική δικαιοσύνης. Θα ήθελα επίσης να σας πω για τις επισκέψεις μου στα κέντρα μετανάστευσης, στα hot spot, τους καταβλισμούς ε, των μεταναστών στην Τουρκία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Κάποια κέντρα και καταφύγια σε άλλα χώρες που συμμετέχουν. Ως αποτέλεσμα, το γραφείο μου δημοσίευσε μια έκθεση που φέρει τον τίτλο «Από την υποδοχή στην αναγνώριση, εντοπισμός και προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων». Ήδη λέμε λοιπόν σε αυτή την έκθεση ότι τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά. Ο στόχος μας είναι η βελτιωμένη αναγνώριση, εντοπισμός και προστασία των δυτικών θυμάτων ανάμεσα στους μετανάστες και κάνουμε λόγο επίσης για το ρόλο και τις ευθύνες των διαφόρων φορέων Είναι, αλήθεια. Είναι σαφές ότι χρειάζεται να υπάρχει μια αναρμονισμένη αρχιτεκτονική για την αντιμετώπιση των αναγκών, καθώς και η άμβληση της, εμπορία, της πιθανότητας εμπορίας, ε, άσχετα από το καθεστώς των μεταναστών ή τις αιτήσει τους. Το αν δεν μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό, μπορεί να οι ότι αυτοί οι άνθρωποι να πέσουν τελικά θύματα των διακινητών και των εμπόρων. Οι εγκληματικές δραστηριότητες ανθίζουν και ε, πολύ δεξιοτεχνικά ε, παρακάμπτουν τις νομοθεσίες. Χρειάζεται ίσως ένας μηχανισμός συντονισμού από όλες τους οργανισμούς που ασχολούνται με αυτά τα θέματα που να, διευκολύνουν, να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, να βοηθήσει και να μπορούν να βοηθήσουν τα θύματα ε, καταλήλως. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα πρέπει να ε, διέπεται από πρωτόκολλα και κατευθυντήρες γραμμές σε κεντρικό και το ε, περιφερειακό επίπεδο που θα δίνει σαφείς ρόλους για όλους τους φορείς, δηλαδή συγκεκριμένο ρόλο για το κάθε ένα φορέα, είτε είναι υποδοχής είτε είναι προστασίας και φυσικά απόλυτη συνεργασία ανάμεσα στα εισαγγελικά γραφεία, τις αρχές μετανάστευσης και τις ειδικευμένε ΜΚΟ που εργάζονται κατά της εμπορίας. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να ε, τυποποιηθούν ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά. Στην Ελλάδα, εργαζόμενοι με τις αρχές, ε, μάλλον, συγγνώμη, ε, μια τέτοια συνεργασία θα αυξήσει τη δυνατότητα συνεργασίας και με τις αρχές του κάθε κράτους μέλους, τόσο για την επιβολή της νομοθεσίας, όσο και για την ε, προστασία και πρόληψη. θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και στα παιδιά. Έχουμε κατευθυντήριες γραμμές ειδικά εκεί που πρέπει να δοθεί η έμφαση. Έχει με, ήδη πριν 10 χρόνια μιλήσει για αυτά τα θέματα και ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ε, όπως είπαμε στην μετανάστευση. Επιτρέψτε μου να περιγράψω τις βασικές συστάσεις ε, τον ε, των οποίων εργαζόμαστε τα κράτη, παρότι έχουν νομική υποχρέωση να προστατεύουν τα θύματα της ε, εμπορίας ανθρώπων, ε, και υπάρχει και σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη δημιουργία ενός μηχανισμού εντοπισμού και προστασίας και βοήθειας στα θύματα το, της εμπορίας, ε, η Οδηγία 2011 του 36, όπου λέει ότι τα θύματα θα προστατεύονται κατά της θυματοποίησης όταν ε, αυτή συμβαίνει, όταν ε, το, μαρτυρούν στα δικαστήρια. Θα πρέπει λοιπόν να κράτη-μέλη να φτιάξουν το κατάλληλο νομικό και διοικητικό πλαίσιο για να απαγορεύσουν και να τιμωρήσουν τέτοιες ενέργειες. Ε, οι εθνικές νομοθεσίες λοιπόν θα πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να εξασφαλίσουν ότι από τη στιγμή που υπάρχει βάση ώστε να πιστεύει κάποιος ότι ε, είναι θύμα ε, εμπορίας τότε θα πρέπει να τους δίνεται μια περίοδος 30 ημερών για ανά, και όπου οι ε, διαταγές περί έκδοσης να μην μπορούν να εφαρμοστούν. Επιπλέον, ε, καλύτερος εντοπισμός συχνά γίνεται μέσω της καλύτερης συλλογής ε, δεδομένων για να μπορούν δηλαδή οι άνθρωποι που φτάνουν στα κέντρα υποδοχής ε, να δίνουν συγκεκριμένα στοιχεία, να έχουμε εθνική βάση δεδομένων κάθε φορά και για τα θύματα εμπορίας. Μια λειτουργική τέτοια βάση δεδομένων θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει όλες τις πιθανές παρεμβάσεις όλων των αρμόδιων φορέων και στο πλαίσιο ποινικών ερευνών. Ε, και αυτό έτσι θα μπορέσει να διευκολύνει μια μεμονωμένη προσέγγιση, μάλλον ατομική προσέγγιση για τα θύματα, καθώς και να εντοπίσει ε, τις εθνικές απαντήσεις ε, κατά της ε, εμπορίας. Η πρόσφατη νομοθεσία 47 κάθετος 2017 προσφέρει μια συνολική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των αναγκών των ασυνόδευτων ανηλίκων. Επιπλέον δικλείδες θα πρέπει να θεσπιστούν ώστε να εξασφαλίσουν ε, ότι δεν θα εξαφανιστεί ένας μη συνοδευόμενος ανήλικος αφού έχει μεταφερθεί σε κάποιο ειδικευμένο ε, κέντρο υποδοχής ε, προστασία των παιδιών που πέφτουν θύματα εμπορίας σημαίνει αρχική υποδοχή ώστε να φτιαχτεί το εμπιστοσύνη και να ε, πλαισιωθούν οι σχέσεις ε, του παιδιού με τις αρχές. Αξιότιμοι κύριοι Προβουλευτές, καλωσορίζω τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιγράφονται στην ανακοίνωση της Κομισιόν του 2017 ώστε να επιτείνει τις προσπάθειες κατά της εμπορίας των ανθρώπων. Επίσης, να συγχαρώ την Κομισιόν για την πρόσφατη υπογραφή κοινή δήλωση κατά της εμπορίας ε, που θέλει να αυξήσει το συντονισμό και θα ήθελα να σας καλέσω να σκεφτείτε τις συστάσεις της υπηρεσίας μου στην πρόσφατη μας έκθεση περί μετανάστευσης και προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία με τις διάφορες υπηρεσίες ε, του γραφείου μας με τις ε, διάφορες υπηρεσίες της ε, Κομισιόν, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πιο ευαίσθητη προσέγγιση στην καταπολέμηση του εμπορίου των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία, στον κύριο Γιλούκου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Προστασίας των Ανηλίκων. Europol. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι που με προσκαλέσατε εδώ να έρθω να συνεισφέρω κι εγώ στη συζήτηση για αυτό το σοβαρό θέμα. Εκπροσωπώ τη Europol, λοιπόν, είναι ο οργανισμός που προσπαθεί να στηρίξει τις χώρες μέλη στις διερευνήσεις που γίνονται για σοβαρά εγκλήματα. Και γι' αυτό εγώ θα παρουσιάσω τα θέματα από την οπτική γωνία της πρόληψης και της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος. Έχουν αυξηθεί πολύ τα εγκλήματα αυτά. Το 2013 είχαμε 3.600 περιπτώσεις οργανωμένου εγκλήματος, ενώ το 2016 ήμασταν ήδη στις 5.000. Το 2017, τους πρώτους μήνες του 2018, είδαμε ότι το οργανωμένο έγκλημα διασυνοριακά συνεχίζει να αυξάνεται. Ε, οι κύριοι τομεί όπου δρά το οργανωμένο έγκλημα είναι είτε η λαθροδιακίνηση μετανοστών, τα ναρκωτικά ε, και η εμπορία ανθρώπων. Βλέπουμε ότι αυξάνεται λοιπόν το οργανωμένο έγκλημα και έχουμε να κάνουμε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό που είναι σαφέ πάντω είναι ότι το εμπόριο ανθρώπων αποτελεί μέρος του οργανωμένου αυτού εγκλήματος. Αλλά όχι μόνο. Και τα ναρκωτικά. Απασχολούν πολύ τη Europol. Η εμπορία ανθρώπων όμως αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος το 2018 με 2021. Η Europol βοηθάει τις χώρες μέλη να θέσουν σε εφαρμογή διάφορες δράσεις για την καταπολέμηση αυτού του οργανωμένου εγκλήματος. Υπάρχει ένα ειδικό κέντρο στη Europol που στηρίζει τις χώρες μέλη στη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων ε, οργανωμένων που έχουν να κάνουν με την εμπορία ανθρώπων. Ε, συλλέγουμε στοιχεία, κάνουμε μελέτες και επίσης προσφέρουμε και αναλυτικές δράσεις στήριξης των ε, χωρών μελών, πιο συγκεκριμένα για το θέμα της διερεύνησης εγκλημάτων που έχουν να κάνουν με την εμπορία ανθρώπων. Στόχος της Europol βέβαια είναι να διασφαλίσει αποτελεσματική διερεύνηση κάθε εγκλήματος που έχει να κάνει με την ανθρώπινη εκμετάλλευση. Δίνουμε ιδιαίτερη ε, σημασία επίσης σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την εμπορία ανθρώπων, κατασχέσεις, ε, διώξεις, βασινόμου κλπ. Η Europol με την Eurojust έχουν εκτιμήσει ότι τα αποτελέσματα που έχουμε είναι λιγότερο από 2% που καταλήγουν δηλαδή σε ποινική δίωξη. Βέβαια, οι ευκαιρίες είναι πολλές για το οργανωμένο έγκλημα και για αυτούς που ασχολούνται με την εμπορία ανθρώπων. Εννοείται επίσης ότι η Europol επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο θέμα της εμπορίας ανθρώπων με βάλωτα θύματα, ανήλικες για παράδειγμα. Το 2017 είχαμε 4.634 ε, επιχειρησιακά μηνύματα. Στηρίζουμε τις χώρες μέλη για 1.063 ε, περιπτώσεις ερευνών 5.629 θύματα και 8.445 υπόπτους εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια των ερευνών αυτών. Στηρίξαμε τις χώρες μέλη σε έρευνες για 52 περιπτώσεις ύψης της προτεραιότητας. Περιπτώσεις δηλαδή που είχαν να κάνουν με υψηλού επίπεδου εγκληματικές οργανώσεις. Βοηθούμε επίσης τις χώρες μέλη στις έρευνες στηρίζουμε επιτόπου, δηλαδή συνεργαζόμαστε με τις αρχές των χωρών μελών επιτόπου, αλλά και με τα διάφορα στρατηγία, όπου προσφέρουμε τεχνική στήριξη αλλά και οικονομική για τις έρευνες. Η Europol προσφέρει στις χώρες μέλη επίσης και μελέτες που έχουν να κάνουν με την εμπορία ανθρώπων. Βοηθούμε συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις χώρες μέλη προκειμένου να σχεδιάσουν τις δραστηριότητές τους για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Το 2017 λοιπόν 61% των θυμάτων που εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες, οποίες συμμετείχε και η Europol, ήταν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. 14% ήταν από μη ευρωπαϊκές χώρες, ε, Νιγηρία και Κίνα κυρίως. 25% ήταν από άλλες εθνικότητες που δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Το 2017, 87% των θυμάτων που εντοπίστηκαν ήταν ενήλικες και 4% ήταν ανήλικες. Οι ηλικίες του 9% δεν είναι γνωστές. Πάντα πρόκειτο για εμπορία ανθρώπων από το οργανωμένο έγκλημα. Θέλουμε επίσης να στηρίξουμε τις αρχές των χωρών μελών προκειμένου να εντοπίσουν και την εμπορία παιδιών και να την αντιμετωπίσουν. Τώρα, το θέμα του φίλου. 75% των θυμάτων ήταν ε, θηλυκού γένους. Και κυρίως επρόκειτο για σεξουαλική εκμετάλλευση. Ένα παράδειγμα ερευνών που στήριξε η Europol ξεκίνησε το 2017 και οι σχετικές έρευνες έκλεισαν το 2018. Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νιγηρία ήταν οι χώρες που συμμετείχαν. Διαλύθηκε το οργανωμένο έγκλημα της Νιγηρίας, 90% ε, των υπευθύνων συνελήφθη. Συμπεράσματα. Βάσει των ε, δραστηριοτήτων της Europol. Η εμπορία ανθρώπων σίγουρα αποτελεί κατηγορία του οργανωμένου εγκλήματος. Τα θύματα είναι κυρίως γυναίκες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως πρόκειται για την σεξουαλική εκμετάλλευση. Βλέπουμε όμως εκμετάλλευση και στον τομέα της εργασίας. Η εμπορία ανθρώπων συνδέεται και με τρίτες χώρες, Νιγηρία κυρίως και την Κίνα. Οι μετανάστες που λαθροδιακινούνται προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς και είναι ευάλωτοι στην εκμετάλλευση. Οι χώρες μέλη θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τη βάση δεδομένων της Europol για να μπορούν να ταλάσσουν στοιχεία μεταξύ τους όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα και η Europol για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις και να στηρίζει τις έρευνες τέτοιων οργανωμένων εγκλημάτων χρειάζεται τη στήριξη των χωρών μελών. Θέλουμε κατάλληλους πόρους για να μπορούμε να στηρίζουμε αυτές τις έρευνες. και να βοηθούμε τις αρχές οι οποίες από μόνες τους δυσκολεύονται να τα καταφέρουν. Επίσης πρέπει να υπάρχει νομική δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με τρίτες χώρες όπου το οργανωμένο έγκλημα, και εμπορία ανθρώπων, είναι παρόν φαινόμενο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Λούκου. τώρα το λόγο έχει η κυρία Άννα Χέντε. Παρακαλώ, από την Επιτροπή Γυναικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω σήμερα εδώ και να μοιραστώ τις σκέψεις μου σχετικά με το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων. Είναι η τρίτη μου θητεία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι ένα πληρωματικό μέλος της Επιτροπής ε, ΛΥΠΕ, αλλά και τα ε, πλήρε μέλο τη Επιτροπή ε, Γυναικών και Ίσων Δικαιωμάτων. Η εμπορία ανθρώπων είναι μία από τι μεγάλε προτεραιότητε τη προσωπικέ μου και ε, ήμουν εισηγήτρια της έκθεσης για την εμπορία ανθρώπων, η οποία ήταν ορόσημο στη, στο έργο της Ένωσης για την καταπολέμησή της. Το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων δυστυχώς αυξάνεται παρά τις προσπάθειες που καταβάλουμε όλοι και είναι ε, πολύ ταχεία η αύξησή του στην ε, παράνομη πλευρά της αγοράς. Η εμπορία ανθρώπων αφορά κυρίως γυναίκες και παιδιά που έχουν κάποιο μεταναστευτικό ε, παρελθόν και υπάρχει η μένη αντίστοιχη οδηγία, όμως το θέμα είναι να εφαρμοστεί σωστά. Η οδηγία πολύ συγκεκριμένα στο άρθρο 1 αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πτυχές της καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι όταν εγκρίθηκε η οδηγία γνωρίζαμε ότι οι γυναίκες και οι άνδρες υπόκειται σε διαφορετικό είδος εμπορίας. Όμως οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν το, ε, το μεγαλύτερο ποσοστό των θυμάτων, 76% ε, των γυναικών χαρακτηριστικά. Χρειάζονται λοιπόν μέτρα προστασία για τα παιδιά και τα υπόλοιπα θύματα τη εμπορία ανθρώπων και τα θύματα θα πρέπει να απολαμβάνουν ε, συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Μία από τις πτυχές της οδηγίας είναι η καταπολέμηση της ζήτησης, που είναι και η βάση της εκμετάλλευσης. Ένας τρόπος ε, αντιμετώπισης είναι να ακολουθήσουμε τη ροή του χρήματος, ε, διότι η εμπορία ανθρώπων ε, λαμβάνει χώρα ακριβώς επειδή υπάρχει ζήτηση, υπάρχει αγορά αυτών των υπηρεσιών που προσφέρουν τα θύματα. Και ένα αρκετά αμφιλεγόμενο στοιχείο είναι η ε, ποινικοποίηση των ε, αγοραστών, των πελατών, των θυμάτων ε, εκμετάλλευσης. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ευαισθητοποίηση. Πρέπει να υπάρχει αρκετή ενημέρωση, είτε, είναι σε, είτε η εκμετάλλευση λαμβάνει χώρα σε οικουσανοχής, είτε σε χωράφια. Χρειάζεται λοιπόν να κινητοποιηθούν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Είναι απαράδεκτη η στάση μας και δείχνει την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάληψη δράσης. Δείχνει ότι εν μέρη συνενεί σε αυτήν την ε, κατάφορη ε, παραβίαση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει έντονα και αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Και μπορούν ε, να γίνουν πολλά, χρειάζεται να γίνουν πολλά, ιδιαίτερα στο πλαίσιο πλαίσιο της μετανάστευσης. Χρειάζεται να γίνει ένα σαφής διαχωρισμός που συχνά αγνοούμε. Η διακίνηση και η εμπορία ανθρώπων είναι άλλα πράγματα. Ε, ακόμα και αξιωματούχοι υψηλόβαθμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν αυτό το λάθος και πολλές φορές ε, σκέφτομαι πως ίσως να είναι σκεμμένα όταν ε, διακινούνται άνθρωποι είναι ένα πράγμα, όμως η, εμπορία, η διακίνηση με σκοπό την εμπορία είναι κάτι τελείως διαφορετικό το οποίο λαμβάνει ε, χώρα υπό την απειλή βίας ή σωματικής ή άλλων μορφών ε, μετά από απαγωγές, μετά από ψευδείς υποσχέσεις, από κατάχρηση εξουσίας ή εκμετάλλευση του ευάλωτου χαρακτήρα και της θέσης των θυμάτων. Όλα αυτά οδηγούν στην εμπορία ανθρώπων. Γι' αυτό αν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς πρέπει να διαχωρίσουμε με σαφήνεια την ε, διακίνηση από την εμπορία. Ένας από τους ε, τρόπους ε, αντιμετώπισης είναι η βελτίωση του συστήματος ασύλου και η βελτίωση της προστασίας των παιδιών. Το σύστημα ασύλου έχει δημιουργηθεί και έχει προσαρμοστεί για άνδρες. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι ένας νόμιμος τρόπος αίτησης ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά, χωρίς αυτό, οι μετανάστες θα αναγκαστούν να καταφύγουν στα χέρια των ε, διακινητών και θα πέσουν έτσι θύματα εκμετάλλευσης, θύματα εμπορίας. Χρειάζεται να προσέξουμε ε, για το θέμα της οικογενειακής επανένωσης και ξέρω πως αυτό δεν είναι κάτι που θέλουν να συζητήσουν τα κράτη-μέλη, όμως είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Υπάρχουν γυναίκες και παιδιά ε, που είναι ευάλωτα κινδυνεύουν να πέσουν θύματα εμπορία ανθρώπων και είναι πολύ σημαντικό να χορηγείται άσυλο σε αυτούς ή να έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν άσυλο. Όλοι οι τον άσυλο πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εξετάζει την υπόθεσή του ενώπιον ε, δικαστηρίου. Και από το 2016 παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση τη εμπορία ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν κάνω έκκληση στον Επίτροπο Αβραμόπουλο αλλά και σε όλη την Επιτροπή να αντιμετωπίσουν την τεράστια πρόκληση αυτή. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα για να μείνουμε αμέτωχοι και άπραγοι. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν θέλω να ρωτήσω αν κάποιος από τους βουλευτές που είναι παρόντες θέλει να θέσει ερωτήσεις, ε, Μπάρμπαρα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που έφτασα καθυστερημένα στην ακρόαση, ιδιαίτερα που δεν... Ε, άκουσα την παρέμβαση για τα θύματα εμπορίας από την Ιγυρία ε, στην Ιταλία. Θα ήθελα να, να μπορέσω να ακούσω την ε, γνώμη σας για τη νέα μεταναστευτική πολιτική της Ιταλικής κυβέρνησης. Ε, θέλω να μιλήσω όμως για την ομιλία που έκανε η κυρία Μύρια Βασιλιάδου για τις προόδους που έχει σημειώσει η Κομισιόν ε, σε, την, σε αυτό το πεδίο που όντως συμφωνώ για, σε μεγάλο βαθμό αλλά υπάρχει ένα σημείο σημαντικό που θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση και αυτό είναι πώς συνδυάζεται η στάση της Κομισιόν που εσείς θεωρείτε θετική για την εμπορία και την υποχρεωτική δουλεία ε, πώς συνδυάζεται με την πολιτική της Ένωσης ε, όσον αφορά την εξωτερήκευση της πολιτικής του ασύλου. Γνωρίζουμε ήδη πια από το σχέδιο συμφωνίας ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι θα υπάρξει αύξηση της χρηματοδότησης προς τη Λιβύη και προς μια ολόκληρη σειρά χωρών που δεν είναι σίγουρες ασφαλής όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη Λιβύη συγκεκριμένα ξέρουμε ότι υπάρχει, ε, ότι υπάρχει δουλεία. Δουλεία των μεταναστών. Και γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτό που πολύ σωστά είπε και η Άννα Χέντ, το εμπόριο δηλαδή που γίνεται χωρίς ε, βέβαια συνένεση του θύματος. Στα κοινωνικά ζητήματα ιστορικά ε, εφευρέθηκαν τα συνδικάτα. Όμως για το θέμα των μεταναστών επιτόπου ποιοι είναι, εν γέννη είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και εμείς ε, παρατηρούμε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μια σταδιακή εγκληματοποίηση των ΜΚΟ, δηλαδή γίνεται συνέχεια μια προσπάθεια μαύρωσης ε, των προσπαθειών. Ε, θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό. Συγγνώμη Πρόεδρε, μακρηγόρησα, με ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Στις, 12.30 οι διερμηνείς πρέπει να σταματήσουν την εργασία τους, οπότε γι' αυτό θα δώσω μέσα το λόγο στην κυρία Βασιλιάδου, αφού σε εκείνη απευθύνατε την ερώτησή σας και στους υπολείπους αργότερα αν θελήσουν να κάνουν κάποιο σχόλιο. Παρακαλώ, κύριε Βασιλιάδου. Ναι, η κυρία από την ΜΚΟ. Όχι, δεν θέλω να θέσω ερώτηση. Όταν θα ολοκληρώσει η κυρία Βασιλιάδου, θέλω να απαντήσω με δύο λόγια στο ερώτημα που μου τέθηκε για την Ιταλία. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ στο Ευρωκοινοβούλιο γιατί για να σας πω ειλικρινά, ε, για να είμαι ειλικρινής, χωρίς το Κοινοβούλιο δεν θα είχαμε μια τόσο ισχυρή ε, διάσταση στο φύλλο στην ε, δουλειά μας για τη μετανάστευση και αυτό γίνεται χάρη στη δικά σας ψηφίσματα και την επιμονή σας. Ε, στην εργασία σας. Για το ερώτημά σας, αυτό που προσπάθησα να πω στην αρχή είναι ότι τα δύο τρίτα των θυμάτων είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν προσπαθώ να αποφύγω την ε, ερώτησή σας, απλώς πρέπει να πω δυστυχώς οι ρίζες του προβλήματος, ο λόγος για τον οποίο υπάρχει εμπόριο ανθρώπων είναι ε, ακριβώς τα λεφτά αστρονομικά κέρδη στην Ευρώπη, όπως είδαμε και από τον συνάδελφο από την Europol, και όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και επειδή ο κόσμος χρησιμοποιεί αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρουν αυτά τα θύματα. Οπότε ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται, όλες αυτές οι γυναίκες, κορίτσια και κάποιες φορές δεκάχρονα κοριτσάκια ή ακόμα και μικρότερα στην ηλικία που έρχονται στην Ευρώπη, διερωτώ αν δεν υπήρχε αγορά, αν δεν υπήρχε κέρδος, αν θα ήμασταν εδώ να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μήπως λοιπόν η πηγή του προβλήματος και η πραγματική δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και η πρόκληση, όπως είπε και η Άννα Χέντ, δεν είναι μήπως αυτό που πρέπει να σταματήσουμε, δηλαδή τη ζήτηση. Και γι' αυτό και ακριβώς επιμένω από την άποψη της, ε, της Κομισιόν ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, ποινικοποιήσουν αυτούς που με τη θέλησή τους συμμετέχουν σε αυτό το έγκλημα. Με τον ίδιο τρόπο που απαιτούμε πολιτική ασύλου και πολιτική μετανάστευσης, θα πρέπει όπως όλος αυτός ο κόσμος από όλα τα πλευρές του, της εκμετάλλευσης που εδώ, εν πάση περιπτώσει, εστιάζουμε στα παιδιά και στις γυναίκες, επιτέλους δόξα σε Θεός, επιτέλους ασχολούμαστε συγκεκριμένα με γυναίκε και παιδιά, να διερωτηθούμε τι συνέβη με όλους αυτούς που έχουν εκμεταλλευτεί γυναίκες και κορίτσια. Είναι εύκολο να εστιάσουμε στα παιδιά γιατί μας κάνει να αισθανόμαστε πιο άνετα. Αλλά η πλειοψηφία και το ακούμε από το, από το Europol και το πιστεύουμε 100% είναι γυναίκες. Και είτε είσαι 80 είτε είσαι 8 χρονών παραμένει το, η πληγή όταν έχεις βιαστεί, έχεις βιαστεί. Τελείωσε. Όταν βλέπουμε ένα κορίτσι, ένα, ένα κοριτσάκι στη, μέσα του χειμώνα στο δρόμο, έξω στο δρόμο, ας πούμε θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα σας στη Ρώμη, στην Ιταλία. Ένα κοριτσάκι μη γυμνό. Ξέρω ότι εσείς θα ρωτούσατε, τι μπορώ να κάνω, πώς να σε βοηθήσω. Πεινάς ή μπορείς να ρωτήσεις πόσο πάει. Πέντε ευρώ σου φτάνουν. Τι θα κάνουμε λοιπόν γι' αυτό το 5 ευρώ. Ποιος το δίνει και τι θα τον κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο που θέτει αυτή την ερώτηση. Και για τη ΜΚΟ είμαι πολύ περήφανη γιατί η Κομισιόν έχει μια πλατφόρμα ε, civil Society, Κοινωνία των πολιτών, πάνω από 400 ε, οργανώσεις, πολλές από την Ιταλία. Δύο φορές το χρόνο ε, συγκεντρωνόμαστε στον ίδιο χώρο, αλλά έχουμε επαφές ολόκληρο το χρόνο. Τα 52% των χρημάτων που έχουμε για την καταπολέμηση της εμπορίας πηγαίνει στις ΣΜΚΙΟ και ενημερώνουμε συνέχεια για να μπορούν να σχολιάσουν, να συνεργαστούν μαζί μας και περιμένουμε από κοινού σχόλια για το τη δεύτερη έκθεση πρόοδου που σύμφωνα με την οδηγία προετοιμάζεται από το συντονιστή για την προσπάθεια κατά της ε, ε, εμπορίας. Ε, προωθούμε λοιπόν τις συμβολές και από τις ΜΚΟ. Εκτός από το συντονισμό ανάμεσα στα μέλη. Θα έχουμε έκθεση στα τέλη του χρόνου και είμαι ευτυχής που βλέπω τη συμμετοχή των ΜΚΟ σε όλα αυτά και στη σημερινή σύσκεψη. Ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω αν κάποιος άλλος από τους ομιλητές θέλει να πει κάτι, να απαντήσει κάτι. Μια σύντομη ε, παρέμβαση σε σχέση με το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Συμφωνώ ότι η κατάσταση Ε, ενώ οι ίδιες οι ΜΚΟ ε, λένε ότι περιορίζεται ο χώρος δράσης τους. Ο ΑΣΕ εργάζεται και είμαστε πάντοτε συνεργαζόμαστε πάντοτε με τις ΜΚΟ που είναι πολύ δραστήριες σε όλες μας τις ε, δικές μας δράσεις και προσπάθειες. και οι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει θα πρέπει να βοηθήσουν στι μη κυβερνητικέ να βελτιώσουν τη χρηματοδότηση και να του δώσουν πρόσβαση. Let me just, um, um it's Κοιτάξτε, τώρα είναι 12.30. Οι διερμηνείς τελείωσαν την, ε, το χρόνο εργασίας τους, οπότε για τις τελευταίες ε, αυτές παρεμβάσεις θα σας παρακαλέσω να τις κάνετε στα αγγλικά και να είστε και σύντομοι. Uh, from Europol's point of view, uh, we would like to underline that both uh, focusing on supply of illegal services and commodities and